Good morning, everybody. Καλημέρα σε όλους. Now, in time. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς, μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερησίας διάταξης ως ε, τροποποιήθηκε. Ωραία. Περνάμε στο δεύτερο σημείο. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 18ης και 19ης Απριλίου και της 30ης Μαΐου είναι στα έγγραφά σας. Υπάρχει διερμηνία σήμερα σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Καλημέρα την ελληνική καμπίνα. Βεβαίως ε, η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά μέσω web streaming και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών της 20 Ιουνίου, ε, σας έχουν αποσταλεί οι αποφάσεις της 23 Ιουνίου. Εγκρίνονται επισήμως, δεδομένου ότι δεν είχαμε ενστάσεις μέχρι την προθεσμία της 28 Ιουνίου του 2016. Με εξαίρεση ένα αίτημα του κυρίου Μαλτέζε, ε, το οποίο έχει προσθεθεί στα διάφορα και ενημερώθηκαν ε, γι' αυτό όλα τα μέλη της Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 1η Ιουλίου. Νομίζω τώρα μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Έχουμε την πολύ σημαντική έκθεση για τη στρατηγική για την νεολαία 2013-2015. Η Εισηγητής ο Ανδρέα Μπόξορ, ο οποίος ε, υπέβαλε το σχέδιο έκθεσής του στις 19 Απριλίου. Να σας υπενθυμίσω ότι οι προθεσμίες ήταν 25 ε, Απριλίου για τις τροπολογίες. Υπευλήθησαν 224 τροπολογίες, 16 συμβαστικές τροπολογίες και έχουμε και γνωμοδότηση από την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα είχαμε 19 τροπολογίες από την Επιτροπή προπολογισμών. Ε, θέλει να πει κάτι η συγγήτρια ή μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην υποφορία. Όχι, σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά σας και τους κοιόδης συγγητές και τη γραμματεία βεβαίως να ευχαριστήσουμε και να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχετε κάρτα. Εντάξει. Περιμένουμε. Περιμένω η ψηφοφορία είναι ανοιχτή. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, έχουμε ισοψηφία γι' αυτό. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην απασχόληση 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα τη ψηφοφορίας. απορρίπτεται με την ίδια ισοψηφία όπως και πριν. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά να το πολιτεύσουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 80 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. «81 κατά τμήματα» ζήτησε η φιλελεύθερη. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ υπέρ Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα 84 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλε 3 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την έμπλη 3. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Να με εμπιστεύεστε. Έμπλη 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 91 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ,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 Ε, Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε, αλλά για μένα είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία για την έμπλε νέα. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 113 και 117 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται.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 εγκρίνεται. 135 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην έμπλα 11 στην επόμενη σελίδα, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 της εισηγήτριας και 145 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 148 υπέρ, κατά αποχές υπέρ και πάλι κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 150 της ηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ, υπέρ και πάλι, κατά αποχές εγκρίνεται. 152, α, συγγνώμη, πάμε στην έμπλε 10. Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση, είναι σαφές. Έμπλε 10 υπέρ, κατά Υπέρ και πάλι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 χωριστή ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος της φιλελευθέρων. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11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 υπέρ, κατά, αποχές. Συγγνώμη και πάλι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. 100, 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 170 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται κοντ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κοντ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κοντ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κοντ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την κοντ 8. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κόντ 9 Υπέρ. Κατά. αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την κοντ 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κοντ 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17. 172. Υπέρ. Κατά. Υπέρ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ το υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία για την 178. Στο CTC Alde, Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές. Έγκρινεται. Και πάμε στην κοντ 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Έγκρινεται. Κοντ 6. Υπέρ. Κατά αποχές. Έγκρινεται. Έμπλ 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 187. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 12. Ας ελέγξουμε. Για την 187 παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους. Διαφορά. Έμπλη 12. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Έμπλη 17. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Έμπλη 18. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 22. Ζητείτε επαλήθευση για την 18. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμπλη 22. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 23. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 15 υπέρ. Κατά άποχες. Θα ήθελα να το επαληθεύσουμε. Για την κόντ 15 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κόντ 16. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Του εισηγείται. 193, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α, συγγνώμη, η 194, η πρόεδρος, υπέρ Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 201 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 202. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 25 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θα ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι για την έμπλη 28. Παρακαλώ. Τον 28. Περάς πληροφορίας. Εγκρίνεται. Η 209. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 του εισηγητή. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 2.16. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 217. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 219. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 220. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε παρακαλώ την 218 Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η 221 υπέρ κατά άποχες δεν είμαστε σίγουροι. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Ας ελέγξουμε τη 221. Πέρασε. Απορρίπτεται. 223. Του θήτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 224 Καταπίπτει, συγγνώμη, η 224. Επειδή εγκρίθηκε η 218. Και περνάμε λοιπόν στην 222. Κατέπεσε η 24. 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 15 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ ξανά σας παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική δια του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. 20. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 21. Υπέρ, κα, υπέρ, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ε, ενδεχομένως απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την 22 πέρας απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε παρακαλώ την 25 Εγκρίνεται εγκρίθηκε η 42 καταπληκτή 26 λοιπόν. Πάμε στην 26 σε τμήματα. Όπω ε, όπως έτσι η Άλτε. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κάτα. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακάτω το πρώτο τμήμα της 26. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά Απόχε. Ε, μάλλον εγκρίθηκε, αλλά σε ελέγξουμε παρακαλώ την 27. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Η 34 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Ε, Προφύγει τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχέ. Ενδεχομένω να απορρίφθηκε, αλλά ας ξαναψηφίσουμε, ας λεπαληθεύσουμε. Τροπολογία 2. Πέρασε. Τώρα πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 40. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41. Α, Αποσύρθηκε η 43 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2 υπέρ. Κατά αποχε εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 ναι, να ελέγξουμε, μα θέλετε. Για την 7, παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Οι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της ε, τροποποιημένης έκθεσης. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 6 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον συνάδελφο και φυσικά συγχαρητήρια και προς τους κοιόδες και ευχαριστούμε ιδιαίτερως και την γραμματεία. Περνάμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη έκθεση που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, της Κάμερ Εβερτ. για θέματα που αφορούν ουσιαστικά στην προσβασιμότητα για προϊόντα και υπηρεσίες Το σχέδιο εκθέσεως παρουσιάστηκε στις 30 Μαΐου οι προθεσμίες κατατέθησαν μέχρι τις 7 Ιουνίου, ήσαν 63, δεν ξέρω αν η συγγήτρια θα ήθελε το λόγο. Κυρία Κάμερε Βέρτ. Εν συντομία, να κάνω μια διευκρίνηση. Και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες ε, κάπως έτσι προκλήθηκε μια αλφα σύγχυση για την γνωμοδότηση αυτή. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω με απόλυτη σαφήνεια ότι εγώ με την πρότασή μου δεν έχω σκόπο να ε, εγκαθιδρύσουμε καθεστώς λιγότερης πρόσβασης για τα οπτικοακουστικά περιεχόμενα. Όχι, πιο πολύ πρόσβαση θέλουμε και μάλιστα ε, μέσω τομεακής ε, προσέγγισης στη σχετική οδηγία. Η Σαμπίνε Φερχάιν και εγώ που είμαστε εισηγήτρες για τις αρμόδιες, ε, ε, για αντίστοιχες οδηγίες θέλουμε να τονίσουμε, να τονώσουμε αυτή την πρόσβαση. Τίθεται και το θέμα των δημόσιων και ιδιωτικών σταθμών, το EVU και το AZT και θα πρέπει να κάτσουμε λοιπόν όλοι μαζί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για να βρούμε μια καλύτερη λύση για μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο οπτικοακουστικό υλικό και ελπίζω να αποδεχτούν τις προτάσεις μας ε, και οι ενώσεις ε, αναπήρων για να καταλήξουμε σε μια σωστή πρόταση η οποία θα εξασφαλίσει το, την πρόσβαση αυτή ιδιαιτέρως γιατί στην παρούσα φάση δεν είναι σαφές πότε και αν θα περάσει ο νόμος, η νομοθεσία ε, για το accessibility, για την προσβασιμότητα ε, στο Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα κάνουμε να προωθήσουμε αυτή την νομοθεσία για το οπτικοστικό περιεχόμενο παρά τα όσα θα μπορούσαμε να πετύχουμε στο Accessibility Act. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας όλοι. Παρακολουθήσαμε από κοντά Ακούσαμε τις διάφορες απόψεις και ακούσαμε και την αντίληψη η οποία λέει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα με πιο οργανικό τρόπο. Η Word όμως έχει ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι πολλά μέλη άλλωστε πήραν πάρα πολλά μηνύματα από οργανώσεις αναπήρων σαν παράδειγμα και από ευρωπαϊκά δίκτυα ΑΜΕΑ και υπάρχουν επίσης και πάρα πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν ανήκουν στην Επιτροπή μας ε, και ε, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση τώρα στην αρχή της ψηφοφορίας. Τζούλη, συγγνώμη, αλλά δεν ξανακάνουμε συζήτηση. Η συζήτηση έχει προηγηθεί. Για παρακαλώ κλείσε σύντομα την παρέμβασή σου. Εγώ ζητώ να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Έχω την θέση, την θέση ότι το θέμα δεν έχει συζητηθεί όσο χρειάζεται με τις κοινότητες των ΑΜΕΑ. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρέπει να πείσουμε ακόμα περισσότερο εάν πράγματι νομίζουμε ότι έχουμε βρει μια λύση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε πείσει και δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Κοιτάξτε αυτό πρέπει να τεθεί στην ησυχήτρια βέβαια Νομίζω ότι έχει υπάρξει αλληλεγγύη ε, ως προς αυτό. Νομίζω ότι έχει υπάρξει σωστή επικοινωνία ανάμεσα στην εισηγήτρια και τις οργανώσεις των ΑΜΕΑ. Παρ' όλα αυτά η εισηγήτρια θα μας πει τι γνώμη έχει πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε συμφωνία για να περάσουμε στην ψηφοφορία ανάμεσα σε όλους. Ε, η Σαμπίνα έχει στήσει το λόγο. Από πλευράς του ΕΛΚ θα θέλαμε να μην ε, συμφωνήσουμε με την αναβολή που προτείνεται. Νομίζω ότι και πριν από την έκθεση αυτή και προηγουμένως έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με οργανώσεις ε, ΑΜΕΑ. Δεν είναι καινούργιο το θέμα. Ήμουν και εισηγήτρια, ήμουν και σκιώδης εισηγήτρια για την οδηγία, για την ε, πρόσβασιμότητα των δημοσίων στους σελίδων και ξέρω ότι το Συμβούλιο θα το να δείξει αυτό σε μεγάλο πρόβλημα αν το θέμα του των οπτικακουστικών μέσων μήνυς, το Accessibility Act. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι για τα άτομα με αναπηρία θα εξυπηρετήσουμε μόνο αν προχωρήσει το θέμα αυτό γρήγορα γρήγορα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι το Accessibility Act ως έχει και ως έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα περάσει έτσι στο Συμβούλιο. Ξέρουμε τι γίνεται και ποια είναι η δημόσια συζήτηση και σε ό,τι αφορά και τα δημόσια website. και δεν ξέρω καν τι θα απομείνει αν δεν ασκηθεί πίεση από πολλές ε, πλευρές και πιστεύω ότι μόνο ε, αν ακολουθήσουμε την οδό που προτείνει η Πέτρα μπορούμε να πετύχουμε κάτι γιατί οι φόβοι ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν ε, μπορώ να πω ότι ανησυχώ, γιατί εγώ σκοπεύω να κάνω πολλά στον τομέα αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει αναβολή. Κοιτάξτε, εμεί εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη και προβλέπαμε την ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ για την ειλικρίνεια την οποία επιδεικνύεται, ε, αλλά πρέπει να πω ότι η οδηγία για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να καταλήξει την διαδικασία της πριν από το Accessibility Act. Εγώ παίρνω πάρα πολύ σοβαρά την διαθεσιμότητα την οποία έχετε επιδείξει όλοι οι συγητές και όδης ε, έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια σε όποια πεδία αυτό είναι εφικτό. Κυρίως στα πλαίσια των συγκεκριμένων άρθρων. Εν πάση περιπτώσει το αίτημα λοιπόν είναι να μείνει μέσα στο συγκεκριμένο αντιμές ε, το άρθρο το οποίο μας αφορά. Ε, νομίζω πρέπει να υπάρξει αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης ε, της παρακολούθησης ε, της αποτελεσματικότητας της πρόσβασης. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθεί η πρόσβαση. Πέρα από το γενικότερο θέμα του Accessibility Act, το θέμα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ειδικές αρχές, ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν την αντιστοίχηση με τις κοινοτικέ προβλέψεις. Πάντως, ε, αυτή στιγμή το Accessibility Act τεθεί επισήμως σε συζήτηση, είναι σαφές ότι θα προσθεθούν επιπλέον θέματα και ίσως εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε τροπολογήσεις της συγκεκριμένης αυτής ε, πρότασης νομικής. Πάντως, σε σχέση με τα ραδιοτηλεοπτικά, είναι σωστό να έχει το θέμα αυτό τη θέση του μέσα στις ρυθμίσεις. Άκουσα τις ανησυχίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία και σας καλώ να ξεκινήσουμε αμέσως. Στο άρθρο 1 λοιπόν, έχω την τροπολογία 36. Ποιοι είναι υπέρ, Κυρία Στέβενς, κοιτάξτε, νόμιζα ότι είχαμε ξεκινήσει την ψηφοφορία. Ένα λεπτό μόνο θα πάρω το λόγο, λέει η κυρία Στίβενς. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, δεν γνωρίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο εδώ, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ έχω έρθει σε επαφή και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με επιχειρήσεις που ασχολούνται με τους ΑΜΕΑ. Έχω έρθει σε επαφή και με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα ΑΜΕΑ. Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά τα οποία μου είπανε, Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στο θέμα του Accessibility Act. Accessibility as well, because audio-visual services... Ιδιαίτερα τώρα με τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες νομίζω ότι ε, εδώ θα πρέπει να θέσουμε το θέμα της προσβασιμότητας έστω και σε ειδικό επίπεδο. Αντίθετα, το Accessibility Act ασχολείται με συγκεκριμένες άλλες ε, ε, με άλλους τομείς. Ίσως να υπάρχει μια μικρή επικάλυψη ανάμεσα στα δύο, αλλά είναι δύο πράγματα τα οποία είναι και τα δύο απαραίτητα ξεχωριστά. αν υπάρχουν σαν παράδειγμα κάποιες εξαιρέσεις για την τηλεόραση. Εκεί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει. Κοιτάξτε, λέει η πρόεδρος, πρέπει να σταματήσετε. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους πριν περάσουν στην ψηφοφορία ότι η ουσία είναι να στηρίξουμε τους άμεα, να έχουν πρόσβαση στα πάντα, χωρίς εξαιρέσεις. Κοιτάξτε, ακριβώς αγαπητοί κυρία Στέβενς, εγώ έκανα μια εξαίρεση και σας έδεσα το λόγο Εκτιμώ ιδιαιτέρως αυτά τα οποία έχετε προσφέρει στη συζήτηση, γνωρίζω και τον ρόλο τον οποίο παίζετε στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω εξ ονόματος των μελών της Επιτροπής ότι ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να είναι πιο απαιτητική, θα πρέπει να είναι πιο έντονη στη διεκδίκηση ε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε εμείς να μεταφερθεί στην ε, οδηγία VMS κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διευκρινίζεται ότι στο άρθρο της οδηγίας καλύπτονται τα πάντα. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μέσα μιας οριζόντιας μορφής όπως είναι το Accessibility Act, αλλά στο εσωτερικό κάθε οδηγίας πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη και για αυτή την κατηγορία. Εγώ ήμουν εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτισμού πάνω στα θέματα αναπηρίας και είχα μιλήσει και στην Ολομέλεια. Ε, ό,τι έχει σχέση λοιπόν με υποτίτλους, ό,τι έχει σχέση ε, με τις ειδικέ ε, γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα στην τηλεόραση, κινηματογράφο, ραδιόφωνο κτλ. Λοιπόν, δεν είναι ε, τώρα όμως ε, ο χρόνος ο σωστός για να γίνει η συζήτηση. Δεν έπρεπε να γίνει η συζήτηση. Είναι όμως τόσο σημαντικό το θέμα που δεν μπορούσαμε να μην πάρουμε το λόγο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. 36 παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές, δεκτή. 3 υπέρ και η 38 ταυτόσημη. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 3 και την 38 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτές. Περνάμε στην 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 6 και 42 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές απερίφη 50 υπέρ κατά αποχές απερίφη 51 υπέρ κατά αποχές απερίφη 52 υπέρ κατά αποχές απερίφη 53 υπέρ κατά αποχές απερίφη 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 67 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 68 υπέρ κατά δεκτή 69 καταπίπτει 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 εισηγητής υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 και 72 ταυτόσημοι. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη προφορική τροπολογία στην 23 που είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές, απερίφθη. 25 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 29 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 30 έχει αποσυρθεί 30 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ε, κατά διέρεση ψήφο στην 33 που ζήτησε το ΕΛΤ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 34 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Το σύνολο. Τώρα ξεκινάμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 10 κατά και 2 αποχές. Η έκθεση γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια στην κυρία Κάμερεβερτ. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την συνολική προσπάθεια. Τώρα, σας παρακαλώ να μείνετε στις θέσεις σας, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο για την Προεδρία. Έρχονται οι Υπουργοί, είναι ήδη εδώ και θα ήθελα να τους καλωσορίσω. Ε, well, ε, please, can you take this? Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. We, we are to start now. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη. Ησυχία παρακαλώ. Τζούλι, Τζούλι, παρακαλώ. Sorry. Thank you to our colleagues and also to... Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους υπολείπους. Λοιπόν, θα μιλήσω Ιταλικά. Φορέστε τα ακουστικό σας και βρείτε και το σωστό κανάλι. Έχετε τη γλώσσα σας. Many languages. And we also are in streaming. Έχουμε διερμηνία σε διάφορες γλώσσες και υπάρχει ζωντανή μετάδοση. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή μας ε, την ε, Σλοβακική Προεδρία και κυρίως ε, τους δύο υπουργούς, τον κύριο Μάρεκ Μάντοριτς, Υπουργό Πολιτισμού και τον κύριο Πέτερ Πλάβκαν, ή Πλάβσκαν, Υπουργό Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας και Αθλητισμού. Ξέρω ότι ήδη ε, είχατε ακρόαση στην Επιτροπή Ήτρα για την έρευνα, επομένω είναι η δεύτερη φορά που μιλάτε ενώπιον μια επιτροπής. Παρ' όλα αυτά, σας καλωσορίζω και του δύο. Θα πω μόνο δύο λόγια, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Να πω ότι συνειδητοποιούμε απολύτω ότι δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη σας Προεδρία, επομένω διπλά ε, να σα ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαστε βέβαιοι ότι η Σλοβακική Προεδρία θα μπορέσει να ερμηνεύσει και τις ευαισθησίες και τα αιτήματα της Επιτροπής Πολιτισμού και του Κοινοβουλίου, διότι αναλάβατε την Προεδρία σε μια πολύ δύσκολη ε, και κρίσιμη συγκυρία της ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά το Brexit και μετά τα όλα θέματα που αφορούν την ανθρωπιστική κρίση και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σε εσωτερικό επίπεδο για την ε, ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Ε, θα ήθελα όμως να μπορέσω να βασιστώ μαζί σας σε επάνω σας και στο Συμβούλιο ε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ακόμα και αυτοί που κόφευαν στις απαιτήσει της ε, παιδείας και του πολιτισμού ε, συνειδητοποιούν λίγο περισσότερο και πρέπει να το δούμε και πολύ συγκεκριμένα ότι αυτοί οι δύο άξονες της πολιτικής, ε, στους οποίους ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο της θεματολόγιο, είναι κεντρική σημασία. Δεν υπάρχει πολιτική ασφάλειας και μετανάστευσης και εξωτερική πολιτική και πολιτική συνεργασίας και πολιτικής ανάπτυξης, εάν δεν στοχεύσουμε στην παιδεία, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και σε έναν ευρωπαϊκό χώρο για την παιδεία και στον πολιτισμό και στα πλαίσια της δημιουργικής ε, ε, βιομηχανίας ε, και ε, στην πολιτιστική κληρονομιά και σε αυτά τα οποία θα συζητήσουμε τόσο λίγου στο VMS αλλά και στα πολιτιστικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά εν γέννη. Θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε λοιπόν και όσον αφορά τον προπολογισμό γιατί φέτος ο προπολογισμό του 2017 είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός για τα προγράμματά μας γι' αυτό και θα θέλαμε στεναρή υποστήριξη από εσά. Να δώσουμε λοιπόν αμέσω το λόγο στον Υπουργό Πολιτισμού, πρώτα στον κύριο Ρεκ Μάνταριτ, ο οποίο θα μιλήσει για 10-12 λεπτά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και τι προτεραιότητε τη Σλοβακική Προεδρία, τα οποία έχουμε δει μεν, αλλά εσεί θα μα τα παρουσιάσετε καλύτερα, και στη συνέχεια στον Υπουργό Παιδεία ε, και κατόπιν θα δώσουμε πρώτα το λόγο. Ε, στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές ε, στη συνέχεια ε, για να θέσουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ Μάνταριτς. Ε, Madam Chair, dear guests, allow me to speak uh, in Slovak language. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μιλήσω σλοβακικά, που είναι και επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιον τη Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για πρώτη φορά απευθύνομαι προς εσάς εξ ονοματό τη Σλοβακική Προεδρία του, του Συμβουλίου. Μία από τι μεγαλύτερε προτεραιότητε τη Σλοβακική προτεραιότητα στο θέμα τη επιτροπή σα είναι και ο έλεγχο τη μεταρρύθμιση ε, τη ε, οδηγία για τα οπτικοστατικά μέσα. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τήρησε το χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή αυτή τη αναθεώρηση και το Μάιο λοιπόν του τρέχοντο έτου μα υπέβαλε τη μια σχετική πρόταση. Και έτσι λοιπόν ε, για πρώτη φορά είχαμε συνομιλίε και με τους άλλους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σημαντική αυτή οδηγία ο οπτικοακουστικός κλάδος έχει ε, τροποποιηθεί πάρα πολύ με δεδομένα και των νέων τεχνολογιών. τη ΦΕΝΤΕΝΕΗ φορείς, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αυτό οδηγεί σε μεγάλες αλλαγές στην αγορά των μέσων και οι παραδοσιακοί πάροχοι όπως είναι οι τηλεοπτικές εταιρείες προσαρμόζονται και αυτές και παρέχουν το περιεχόμενό τους και επιγραμμικά στο διαδίκτυο. Αυτό ασφαλώς ε, οδηγεί σε μεγαλύτερες ε, επιλογές ε, και μεγαλύτερη προσφορά και για τον ε, πελάτη, για τον καταναλωτή. Η παραδοσιακή ιδέα τηλεόριση και τα παραδοσιακά περιεχόμενα δεν διακρίνονται ουσιαστικά από τα σύγχρονα αυτά περιεχόμενα από τον καταναλωτή. Ωστόσο, η ρύθμιση είναι διαφορετικοί και οι διαφορές που υπάρχουν είναι μεγάλες και διαγκώνονται. Ο πελάτη ουσιαστικά δεν κάνει διάκριση μεταξύ των περιεχομένων αυτών, μεταξύ του περιεχομένου που βλέπει στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Και αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνει ότι και γιατί υπόκεινται σε διαφορετικέ ρυθμίσει τα περιεχόμενα αυτά. Τελευταία φορά, δε, οι ρυθμίσεις αυτές ελέγχθησαν και αναθεωρήθηκαν πριν από 10 χρόνια. Ασφαλώς, έκτοτε, όπως σας ανέφερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι λοιπές εξελίξεις ήταν πολλές και γι' αυτό λοιπόν καλούμαστε να ελέγξουμε το πλαίσιο. Αυτό, όπως τόνισε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας στα τέλη του 2014. Και ζητήθηκε επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αθεώρηση. Χαίρομαι δε ιδιαίτερα για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα έλαβε όλα αυτά υπόψη τη. Είμαι ταπεπισμένος ότι έχει γίνει ήδη πολύ σημαντική δουλειά αναφορικά με τα θέματα αυτά και αναφορικά με τους τομεί που αγγίζει η νομοθεσία αυτή. Και θα ήθελα να υποδείξω στο σημείο αυτό την νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή σα. Τα θέματα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και η Σλοβακική Προεδρία έχει ε, ως προτεραιότητα ιδιαίτερος την προστασία των ανηλίκων, μιας και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες καταναλωτών σε ό,τι αφορά τις νέες αυτές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα είναι και μία από τις πιο ευάλωτες ή πιο ευάλωτη ομάδα. Θεωρώ πιστε, ότι η αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει να επιτυχάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των ε, ανηλίκων ανάλογα, ανεξάρτητα από το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. Διοργανώθηκε λοιπόν και μία ένα συνέδριο για την ε, νομοθετική σύγκληση σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων. Και αυτό αποτελεί ένα σημείο κλειδί στην όλη φάση περισυλλογή. Στο συνέδριο θα λάβει χώρα μεταξύ 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 2016 στην Μπρατισλάβα. Η σλοπακική Προεδρία προτίθεται να σημειώσει όσο μεγαλύτερη πρόοδο γίνεται σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των σχετικών διαπραγματεύσεων και ήδη το μήνα αυτό ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας για τα όπτικα ακουστικά και θα συνεχίσουμε εντετικά τις συζήτησεις αυτές μετά το θερινό διάλειμμα. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας που έχει και σπουδαία βιογνωμοσύνη και πολλά χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό και την ίδια στενή συνεργασία έχουμε και με τις Προεδρίες της Μάλτας και της Ολλανδίας. Δεδομένης ε, της περιπλοκότητας των ε, διαπραγματεύσεων αυτών, σκοπεύουμε να καταθέσουμε και μια έκθεση προόδου στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου για την ε, εκπαίδευση, την νεολαία, νεολαία και τον αθλητισμό. Μία άλλη προτεραιότητα στον τομέα της, του πολιτισμού είναι η πρόταση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου προκειμένου το έτος 2018 να ανακηρυχθεί έτος πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσπάθεια που έχει καταβάλει για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής από κοινού με το Συμβούλιο. Είναι τιμή μας το ότι ξεκινούμε τις εργασίες αυτές κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η κοινή πολιτισμική κληρονομιά είναι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα, θεωρεί η Σλοβακία, της προσπάθειας να δοθεί νέα πνοή στι αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης για τους πολίτες σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε σημαντικές οικονομικές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Πιστεύουμε δε ότι η επένδυση στην κληρονομιά μα δεν είναι μια άσκηση κατά την οποία δαπανούμε και εξοδεύουμε χρήματα. Όχι, ουσιαστικά επενδύουμε για το μέλλον και μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο πάρα πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά την προοπτική ανάδειξη του έτου 2018 έτους πολιτισμικής κληρονομιάς, τονίζονται όλες οι ευκαιρίες που θα σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαιρόμαστε που αντιμετωπίζουμε τρεις προκλήσεις στο σημείο αυτό. Την πολιτισμική ε, ποικιλομορφία, τις δημογραφικές αλλαγές και τη βιωσιμότητα. Στο ευρύτερο πλαίσιο θα τονιστούν και οι αξίες της πολιτισμικής ε, ποικιλομορφία και πολυμορφίας της Ευρώπης. Ε και εστιαζόμαστε στην περιφερειακή και εθνική διάσταση σε διάφορα την πολιτισμική κληρονομιά. Πολλά θα είναι τα project, τα τοπικά έργα, τα τοπικά προγράμματα τα οποία θα δανειστούν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Και αυτό θα μπορούσε επίση να αποτελέσει μια τεράστια όθηση για την ε, δημιουργία θέσεων εργασία, καθότι θα υπάρχουν και ευκαιρίε ε, εορτασμών για σε διάφορα μέρη ω τμήμα τη. Ε, Ευρωπαϊκή μα ε, ευαισθητοποίηση και αυτό που υπογραμμίζουμε είναι ότι το 2018 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου ε, Πολέμου και την, την ε, επέτειο 400 ετών της έναρξης του 30ου πολέμου και επίσης τη σύνθηκη της βεσφαλία το 1648. Επίση, από κοινού με το Κοινοβούλιο σκοπεύουμε να συνεργαστούμε και ιδιαίτερω με την Επιτροπή σα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα τη σχετική πρόταση. Μόλι τη λάβουμε, η Σλοβακική Προεδρία θα κάνει το παν δυνατόν για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσει σε επίπεδο Συμβουλίου. Η τελευταία μεγάλη προτεραιότητα στον τομέα της ε, εκπαίδευσης θα είναι η διαμόρφωση των διαπολιτισμικών σχέσεων. Ο πολιτισμός παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο, α, αναντήρητο ρόλο στις σχέσεις τις ευρωπαϊκές. Η Σλοβακική Προεδρία καλωσορίζει λοιπόν την ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Διαπολιτισμικές Σχέσεις και η Προεδρία θεωρεί ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική συμβολή για την, ε, το εσωτερικό αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συγκαταλέγεται λοιπόν αυτό ανάμεσα στις προτεραιότητες μας και θα αναζητηθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η στρατηγική που προτείνεται λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τις αρχές που είχε καθορίσει το Συμβούλιο, για παράδειγμα, στα συμπεράσματά του του 2015, του Συμβουλίου του 2015 για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και σε ό,τι αφορά την ε, συμβολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπη στι ε, παγκόσμιες διαπολιτισμικέ σχέσει. Σκοπεύουμε να θέσουμε το θέμα αυτό και σε σχετικό συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι αγαπητοί ευρωβουλευτέ, και προσβλέπω στι μελλοντικέ μα συζητήσει. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πολύ σημαντικές οι προτεραιότητές σας, συνάδουν και με τις δικές μας τις προτεραιότητες και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά μαζί. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Υπουργό Πλάτκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού. Βάσει και του εθνικού μας προγράμματος, ε, η ε, ανάπτυξη του ταλέντου είναι βασική προτεραιότητα στον τομέα της παιδείας, ε, του αθλητισμού και της νεολαίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στους πολίτες της. Επομένως, ε, σήμερα ως δυναμική κοινωνία πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό. Η Σλοβακική Προεδρία φρονεί ότι η υποστήριξη του ταλέντο είναι ένας τρόπος να δώσουμε μια όθηση στην ανταγωνιστικότητα, να ε, βοηθήσουμε τον ανταγωνισμό και να συνεισφέρουμε στην προσωπική ανάπτυξη του καθενός. Χωρίς αμφιβολία το ταλέντο είναι ο κινητήριος μοχλός ε, της ε, οικονομικής ανάπτυξης επίσης, της αποτελεσματικής οικονομικής ανάπτυξης δε. Όλα αυτά σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής πρωτοβουλίας και της, ε, του θεματολογίου για την νεολαία και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται όχι μόνο για την κυκλοφορία, την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά επίσης ε, δεξιότητες ε, και προσόντα τα οποία απαιτούνται για να συμμετέχει κανείς στη ζωή ως ενεργός πολίτης. μέσω της διαπραγμάτευσης ε, των συστάσεων του Συμβουλίου για την εγγύηση για τις δεξιότητες θα προωθήσουμε τα θέματα αυτά, κυρίως ψηφιακές δεξιότητες, επιχειρηματικές και εγκάρσιες δεξιότητες. Στα πλαίσια του πλαισίου για την ε, νεολαία θα έχουμε συγκρισιμότητα των προσόντων που θα περιλαμβάνουν γνώση, δεξιότητες και αρμοδιότητες οι οποίες απαιτούνται για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, θα επικεντρωθούμε και στην ε, θεματολόγιο για την ανώτατη εκπόδευση και τις ε, ψηφιακές δεξιότητες. Η πολιτική συζήτηση από τους υπουργού για το Συμβούλιο Παιδείας που προβλέπεται για τον Νοέμβριο του 2016 θα ε, έχει ως θέμα ανάπτυξη και υποβοήθηση του ταλέντου. Η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι βασικός ε, ε τομέας της καταπολέμησης του εξτρεμισμού και επομένως πρέπει να υπάρχει συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παιδεία, είτε επίσημη είτε άτυπη παιδεία ε, και φυσικά ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης ε, και κοινωνικών γνώσεων. Αυτό θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη δικλίδα ασφαλείας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και κατά συνέπεια και κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Γνωρίζουμε ότι στον τομέα αυτό υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωση σε πολλά κράτη-μέλη, καθώ επίση και περιθώριο πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ε, ε, σχετικών ενδιαφερομένων μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίο εξτρεμισμό, ε, θα προτείνουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία μεταξύ άλλων θα επισημάνουν και τη σημασία της παιδείας που περιλαμβάνει τους πέντες και την ανάγκη να προσπαθήσουμε να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Τα συμπεράσματα θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν ε, την ε, παιδεία που περιλαμβάνει τους πάντες, ε, ανάπτυξη αγωγής του πολίτη, καθώς επίσης και προώθηση αξιών μέσω της παιδείας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, καθώς επίσης και της υποστήριξης μιας προσαρμοστικής κοινωνίας που περιλαμβάνει τους πάντες και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους νέους. Ε, με βάση τις προκλήσεις ε, που προκύπτουν και από το μεταναστευτικό κύμα θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης της ένταξης ε, των υπηκών τρίτων χωρών το οποίο δημοσιεύθηκε προσφάτως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία στον τομέα της παιδείας, του αθλητισμού και της νεολαίας και του αθλητισμού, συγγνώμη. Ε, θα υπάρχουν ε, οι συνήθεις συναντήσεις με τους γενικούς διευθυντές και μεταξύ των θεμάτων θα περιλαμβάνονται συγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, κυρίως ε, η ανώτατη παιδεία και η σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, αποτελεσματική χρήση των πόρων στην παιδεία, και μία ε, παρακολούθηση της εφαρμογής όλων αυτών από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία και την προώθηση της αριστείας ε, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το βασικό θέμα της Σλοβακικής Προεδρίας ε, θα το αντιμετωπίσουμε στη διάσκεψη Flexit για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του ταλέντου στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Στη διάρκεια αυτής της ε, διάσκεψης θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ταλέντο σε όλους τους τομείς της παιδείας, καθώς επίσης και στην κοινωνία και στις τέχνες. Η διάσκεψη θα επικεντρωθεί στην υποβόθηση και ανάπτυξη του ταλέντου από τρεις άξονες, κυρίως ένταξη, δηλαδή τη δυνατότητα οι διδάσκοντες να ανακαλύψουν, να ε, αναπτύξουν και να υποστηρίξουν το ταλέντο από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ε, ανεξάρτητα από το ε, πού προέρχονται τα παιδιά. Μετά θα επικεντρωθούμε σε ε, άριστους μαθητές και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτύξουν πλήρως το ταλέντο τους ε, τα παιδιά αυτά. Και τρίτον, ε, θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τις ειδικέ δεξιότητες και ταλέντα που έχει το κάθε παιδί για να βοηθήσουμε αυτά τα οποία έχουν ένα χάρισμα και δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το αναπτύξουν καταλήλους. Όσον αφορά την νεολαία, θα εξετάσουμε το ταλέντο από ευρύτερη σκοπιά. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε και να αναπτύξουμε το ταλέντο και τις δυνατότητες των νέων παιδιών μέσω συγκεκριμένη προσέγγισης ε, στην εργασία για τους νέους. Το περιβάλλον εργασίας των νέων θα πρέπει να είναι ελκυστικό, σύγχρονο και να αντακατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων. Ιδάλλως ε, θα υπάρχει μείωση στη δέσμευση και στη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Οι αλλαγές ε, στον τρόπο ζωής ε, των νέων ανθρώπων ε, απαιτούν επίσης και την εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας των νέων, είτε σε διαδικτυακό περιβάλλον, είτε και εκτός διαδικτύου. Η Σλοβακική Προεδρία θα εγκρίνει συμπεράσματα του Συμβουλίου για νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των νέων, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Σε επίπεδο κρατών μελών χρειαζόμαστε με πιο εντατική ανταλλαγή εμπειριών, διότι το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, αλλά δεν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα και επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Πέραν των εγγράφων πολιτικής, ε, συντάσσουμε με την μελλοντική Μαλτέζικη Προεδρία ε, ένα ε, ε, έγγραφο για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Ο τρίτος διαρθρωμένος διάλογος ε, στο τρίο των Προεδριών Ολλανδία, Σλοβακία, Μάλτα έχει ως σύνθημα το έτοιμη για την νεολαία, έτοιμη για την κοινωνία που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε επιτυχή ανάπτυξη των νέων σε μια ποικιλόμορφη Ευρώπη που περιλαμβάνει τους πάντες. Ε, θα γίνει τον Οκτώβριο στην Κόσιτσα και μια σχετική διάσκεψη. Τα αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής ε, θα δοθούν εν είδη συμπεράσματων, θα συζητηθούν στο Συμβούλιο ε, Υπουργών Παιδείων και στη συνέχεια θα έχουμε και συνάντηση Γενικών Διευθυντών για την Νεολαία με ε, κύριο θέμα την υποβοήθηση και την ανάπτυξη του ταλέντου των νέων ανθρώπων. Στην ε, συνεδρίαση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τις προτεραιότητες για τη νέα στρατηγική για την νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα παρουσιάσει και ε, τα ευρήματά της από την ενδιάμεση αναθεώρηση της παρούσας στρατηγικής και η Σλοβακική Προεδρία σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις για τις μελλοντικέ προτεραιότητες και την ε, ε, παρακολούθηση της πολιτικής για την νεολαία μετά από το 2018 θα προσπαθήσουμε να ε, γκρίνουμε μία ε, εγκάρσια προσέγγιση που ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την νεολαία. Η πολιτική για την νεολαία δεν είναι μόνο αρμοδιότητα των Υπουργών Αρμοδίων για την νεολαία. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς και πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν πολύ σημαντικά την ποιότητα της ζωής των νέων ανθρώπων Όσον αφορά τον αθλητισμό, θα επικεντρωθούμε κυρίως στις θετικές πτυχές ε, και επομένως ε, σε συνδυασμό με το ε, πρόγραμμα της Προεδρίας θα πρέπει να δούμε τον αθλητισμό, την αθλητική διπλωματία και τις πολιτικές για την νεολαία. Στον τομέα του αθλητισμού έχουμε ένα κοινό παρονομαστή, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στον αθλητισμό. το θεματολόγιο της Ομάδας Εργασίας για τον Αθλητισμό θα ξεκινήσει συζητήσεις για επίκαιρα θέματα, όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση της εφαρμογής του Δευτέρου Προγράμματος Εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο μέχρι το 2017, καθώς επίσης και την προετοιμασία ενός ε, πιθανού τρίτου σχεδίου για το επόμενο διάστημα. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει σχέση και με τα όσα κάνει η δική σας η Επιτροπή, γιατί εσείς καταρτίζετε έκθεση για την ε, καλύτερη προσέγγιση στην πολιτική για τον αθλητισμό μέσω καλής διακυβέρνησης, Προσβασιμότητα και ακεραιότητας. Οι συνέπειε του αθλητισμού στην προσωπική ανάπτυξη θα είναι το θέμα τη συζήτηση των Υπουργών στο Συμβούλιο για τον Αθλητισμό, όπου θα συζητηθούν θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω έγινε και από το 2004, που ήταν το ευρωπαϊκό Έτο ε, του αθλητισμού. Προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας ε, θα συζητηθούν στη διάρκεια της διάσκεψης ε, εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού την επόμενη εβδομάδα στην Πρατισλάβα με συμμετοχή ε, αρκετών ε, ενδιαφερομένων από τα κράτη-μέλη, εμπειρογνωμόνων από τρίτες χώρες, καθώς επίσης ε, και επιτυχείς αθλητές, Σλοβάκους Ολυμπιονίκες και ούτω καθεξής. Θα έχουμε και μία άτυπη συνεδρίαση των ε, διευθυντών αθλητισμού, όπου θα συζητήσουμε τις βασικές μας προτεραιότητες από κυβερνητική σκοπιά. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο θέμα του ντόπινγκ. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην καταπολέμηση του ντόπινγκ η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενωμένη και δυνατή. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού θα διεξαχθεί επίσης στη διάρκεια της Προεδρίας μας και θα γίνει και μία ε, τελετή έναρξης ε, το Σεπτέμβριο στην Κόσιτσα με συμμετοχή του Επιτρόπου Ναυράστσιτς ε, και καθώς και άλλων διακεκριμένων προσκεκλημένων του τομέα του αθλητισμού. Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση του ε, Συμβουλίου Αθλητισμού θα γίνει 21 και 22 Νοεμβρίου του 2016. Προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία μαζί σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προτεραιότητες που μας παρουσιάσατε, κυρίως τα θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές για τους νέους, ε, για το ταλέντο τους ε, και να πω ότι θα είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λογικά και εγώ στην διάσκεψη για τον αθλητισμό που θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Ε, καταρτίζεται και μία έκθεση του συναδέλφου Τάκουλα για το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική και η πολιτιστική διπλωματία μέσω του αθλητισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, όπω επίση και όλα τα θέματα που αφορούν το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη και την ε, κοινωνική συμμετοχή ατόμων τρίτων ε, χωρών, ε, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει περισσότερο περιθώριο για φοιτητέ, ε, διδάσκοντε και του κόσμο του πολιτισμού. Να δώσω το λόγο στου σε Η κυρία Φερχάγεν, η κυρία Καμερέβερ και ο... Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω εξ τη της ομάδας μου του ΕΛΚ για την παρουσίαση των εργασιών σας για το επόμενο μισό έτος. Ένα θέμα θα ήθελα να θέξω, κύριε Υπουργέ. Αναφέρατε την οδηγία για τα οπτικοακουστικά. Θέλουμε να καταλήξουμε και στη δική μας θέση τον επόμενο, τους επόμενους μήνες από πλευρά της Επιτροπής με το θέμα αυτό και γίνεται μια συζήτηση σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την προσβασιμότητα η Επιτροπή μας ενδεχομένω να θέλει να βγάλει τα το μέσα από την ε, νομοθεσία αυτή. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθεσία που ως σκοπό έχει την ε, επίτευξη προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για, τους, ε, για τα αμαία. Ερωτώ λοιπόν, κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη αυτό το θέμα στις ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά δηλαδή τα απτοκοστικά μέσα και τη συμπερίληψή τους στην ε, νομοθεσία και την προσβασιμότητα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μας υποστηρίζετε λοιπόν και γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η τοποθετησή για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι ε, ιδιαίτερα στο θέμα της οδηγίας για τα οπτοκουστικά θα πρέπει να βρούμε σωστές λύσεις και ιδιαίτερα για τους νέους, προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους στην αγορά. Γιατί είναι πολύ υπάροχοι και είναι πολλές οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται. Για τα θέματα των προγραμμάτων Εράσμους και για τα θέματα του αθλητισμού στο, στους επόμενους μήνες, στους επόμενους έξι μήνες, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα γίνει μια αναθεώρηση και για, από την Επιτροπή μας για την εξέλιξη των προγράμματων αυτών. Το θέμα λοιπόν της απλοποίησης των προγραμμάτων και της ε, μεγαλύτερης και ευκολότερης πρόσβασης στα προγράμματα για τους χρήστες των προγραμμάτων, κατά πόσον ε, παίζει ρόλο για την ε, Προεδρία σας, θα θέλαμε να ξέρουμε. Οπότε συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και των οργανώσεων και των νέων. Ακούμε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκες οι διαδικασίες των θεσμικών οργάνων. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζονται ειδικέ ρυθμίσεις για τις μικρές οργανώσεις. Και τι γίνεται για τα, με τα μέσα για την Ευρώπη, για τους πολίτες. Υπήρξε περικοπή 25%. Και ξεκίνησε πάλι μετά τον Brexit και η όλη η συζήτηση για το πώς θα πρέπει η Ευρώπη να προσεγγίσει τον πολίτη. Η Επιτροπή μας επανελειμμένα έχει ζητήσει να μην γίνονται περικοπές σε τέτοια προγράμματα, γιατί η συνάντηση των ε, ανθρώπων από όλη την Ευρώπη και εκτός από τις δυνατότητες εκπαίδευση και εκτός των ορίων του ερασμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Να συναντιούνται λοιπόν οι πολίτες να συζητούν τα ευρωπαϊκά θέματα πέρα από τα εθνικά σύνορα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς τοποθετήσετε για τα θέματα αυτά. Γιατί σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού υπάρχουν διαρκώ ζητήματα σε ό,τι αφορά και την συνάντηση λοιπόν των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας στην ε, Προεδρία σας. Έχετε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Είναι φιλόδοξη η στόχη που έχετε θέσει για την επεξεργασία όλων των θεμάτων αυτών τα επόμενα, τους επόμενους έξι μήνες. Κάθε επιτυχία σας ευχόμεθα. Και θα ήθελα να περιοριστώ στην ε, οδηγία για τα οπτοακουστικά. Είμαι εισηγήτρια και εγώ, όπως και η Σαμπίνε, και αυτό θα καθορίσει το έργο μας τους επόμενους ε, μήνες. Και γι' αυτό χαίρομαι λοιπόν που έχετε θέσει το θέμα αυτό σε, ως μία από τις προτεραιότητές σας. Και καλό θα ήταν να καταλήξει και το Συμβούλιο σε μία κοινή τοποθέτηση από ό,τι άκουσα συνεργάζεστε στενά και με, την Μαλτέζικη, με τη Μαλτέζικη Προεδρία που θα αναλάβει τα καθήκοντά τη από 1η Ιανουαρίου και προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τη Σλοβακική Προεδρία γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε επισταμένο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρόλα αυτά να καταλήξουμε άμεσα, γρήγορα σε μια λύση, γιατί φυσικά δεν μας περιμένει κανείς και ο χρόνος κυλάει και χρειαζόμαστε λοιπόν μια σωστή, ορθή λύση η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στην ανάγκη του μέλλοντος. Γιατί όπως είπατε, οι διαδικτυακές ή μη υπηρεσίες πλέον δεν διαχωρίζονται καν από πλευρά του καταναλωτή. Ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουν το θέμα των γραμμικών και των μη γραμμικών ε, υπηρεσιών όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι για όλους τους φορείς της αγοράς, το οποίο ελπίζω να αντέξει και σε βάθος δεκαετίας. Το τονίζω αυτό, γιατί αυτό ασφαλώς θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους μας. Πώς θα διαμορφώσουμε μία νομοθεσία η οποία θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές τεχνολογικέ ε, εξελίξει, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι σε πέντε χρόνια να είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο και να είναι πάλι παροχημένη η οδηγία και να χρειάζεται να την ε, ενημερώσουμε και να την εξυγχρονίσουμε εκ νέου. από πλευράς λοιπόν προστασίας του καταναλωτή και των νέων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές της διανομή και κατασκευής οπτικοστικοτικών μέσων και για θέματα πλουραλισμού και επικοινωνία στον κλάδο αυτό στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες θα μπορούν να αντέξουν κάπω στη δοκιμασία του χρόνου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που συνεργάζεστε μαζί μας προς την κατεύθυνση αυτή και όπως σας είπαμε και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια λύση. Για το Erasmus Plus, για το Erasmus Sin. πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αναμφίβολα θα μας απασχολήσει και αυτό στο μέλλον. Η Σαμπίνε Φραχάιν τόνισε ότι πολλοί από τους ε, ενδιαφερόμενους δηλώνουν ότι αυτοί οι στόχοι που έχουμε θέσει και στο Κοινοβούλιο για την καλύτερη προσβασιμότητα, την απλοποίηση, την ε, μεγαλύτερη προβολή προγραμμάτων παλιών όπως το τα Νταβίντς, το Κομένιους, όλα αυτά λοιπόν ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πολλά σημεία μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελεί στόχο μας ε, η συνέχιση αυτού του επιτυχούς προγράμματος με τη σωστή χρηματοδότηση, ενδεχομένως και με πιο πολλούς πόρους από ό,τι είχαμε στην ως τώρα, αλλά κυρίως να φροντίσουμε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε να μας υποστηρίξει το Συμβούλιο. Ίσως όχι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, αλλά τουλάχιστον στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Να πείσουμε το Συμβούλιο ότι ένα τέτοιο σημαντικό πρόγραμμα για τους νέους αλλά και για τους πιο ηλικιωμένους είναι ευκαιρίες για εμπειρίες στο εξωτερικό και ίσως λοιπόν ε, στο σημείο αυτό να ήταν διτεθειμένο το Συμβούλιο να βάλει το χέρι λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. Ευχαριστούμε. κυρία Τρούπελα. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Άκουσα προσεκτικά αυτά τα οποία είπατε ότι θα κάνετε και έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το AVMS. Αναφερθήκατε στο ότι είστε υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων. Μία από τις προτάσεις αυτές είναι η ε, προφύλαξη των ανηλίκων από ρητορικές μίσους ε, κτλ. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν είστε υπέρ της πρότασης αυτής και αν το υποστηρίζετε. Και για το Erasmus Plus. Την προηγούμενη εβδομάδα το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ξεκαθάρισε και είπε ομόφωνα ότι χρειάζεται για τα τρία αυτά προγράμματα αύξηση του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για το Erasmus θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν η Σλοβαγική Προεδρία θα υποστηρίξει την πρόταση για το Erasmus Plus. Και να έλθω σε αυτό που είπε η κυρία Κάμερεβερτ. Πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γερμανίας από όπου προέρχομαι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για το Erasmus και τα διάφορα υποπρογράμματα, παραπονούνται ότι οι αιτήσει είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε μαζί μας για να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα έτσι ώστε οι αιτήσει να μπορεί να συμπληρωθούν ευκολότερα. Ε, επειδή θέλουμε να καλύψουμε πάρα πολλές ομάδες ε, της ε, κοινωνίας, φοβάμαι ότι δημιουργούμε μια μεγάλη δυσθυμία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την αίτησή τους και δεν τους προσελκύουμε στα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν θέλετε να κινηθείτε και προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί θα γίνει μια συζήτηση για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών και χρειάζονται αλλαγές. θα δώσω το λόγο στους υπουργούς και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Μαντάριτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις και τις ερωτήσεις. Ε, να πω στις ε, κυρίες οι οποίες πήραν το λόγο προηγουμένως ότι ειδικά για την οδηγία για τα α, μέσα τα οπτικοακουστικά μέσα ανεξάρτητα από το επίπεδο ποιότητας της οδηγίας οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ ε, γρήγορες και θα ήμασταν ε, ικανοποιημένοι η τρίτη οδηγία να κρατήσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Όπως είπα ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα δυναμικός. Το 2007 δεν ήμασταν σε θέση να προβλέψουμε τις αλλαγές οι οποίες γίνονται σήμερα. Και έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις που η καθεμία από σας έθεσε. θέλουμε να κάνουμε μια διάσκεψη της Προεδρίας για την προστασία των ανηλίκων. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ε, το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τη Σλοβακία, τη Σλοβακική Προεδρία. Για την αναθεώρηση της οδηγίας φυσικά σαν προεδρεύουσα χώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις θέσεις των διαφόρων κρατών μελών Είναι σαφής όμως η ανάγκη για κάποιες ρυθμίσεις στον τομέα αυτό που δεν θα αφορά μόνο στις ε, τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και στις συνολικότερες πλατφόρμες. Εμείς λοιπόν σαν Προεδρεύουσα χώρα είμαστε υπέρ της προθεσμίας πρώτων των ανηλίκων και για τους λόγους τους οποίους προανέφερα γιατί αποτελούν αν θέλετε τη μεγαλύτερη ομάδα θέασης ε, ε, τηλεθέασης και ταυτόχρονα και την πιο ευάλωτη. Σήμερα το πρωί είδα το BBC και είδα μια έρευνα την οποία είχαν κάνει που έλεγε ότι τώρα πια ο κόσμος, είναι ιδιαίτερα, η νέα γενιά δεν βλέπει τόσο τηλεόραση όσο άλλες πλατφόρμες όπως τα πάντα, τα smartphones κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό, λοιπόν δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Τώρα για την κυρία Βερχέγεν και την προσβασιμότητα. Εδώ θα πρέπει να δεχθούμε ότι η οδηγία δεν περιλαμβάνει τα θέματα που έχουν σχέση με την προσβασιμότητα. Το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για το Accessibility Act που περιλαμβάνει τα οπτικοακουστικά. Τα θέματα αυτά ε, είναι σε επίπεδο συζήτηση στην αρμόδια τεχνική ομάδα του Συμβουλίου. Αν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, για, την, ε, για το Accessibility Act πάλι έχουμε κάποιες δυσκολίες για να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις προτάσεις, τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί για τους ΑΜΕΑ. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι θα πρέπει εμείς να συμπεριλάβουμε το θέμα της προσβασιμότητας στην διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας. Ο κύριος Πλάφτσαν έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω τις ερωτήσεις και να δώσω κάποιες κοινέ απαντήσεις και στις τρεις προλαλήσασες. Πράγματι το Erasmus Plus είναι το πιο πετυχημένο πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά στοιχεία χάρη στο πρόγραμμα αυτό, 3 εκατομμύρια νέων έχουν την δυνατότητα να φεύγουν από τις χώρες τους για συγκεκριμένα χρονικά διασήματα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν το πρόγραμμα αυτό για το σύνολο της Ένωσης. Σχετικά τώρα με τις προτάσεις οι οποίες έγιναν για την αύξηση του προϋπολογισμού, φυσικά και είμαστε υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού για τα προγράμματα αυτά. Γιατί όπως είπα, είναι ιδιαίτερος επιτυχή. Σχετικά τώρα με την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν 7 επιμέρους προγράμματα στην ουσία μέσα στο Erasmus Plus και υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία και χρησιμοποιούνται 16 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις καταθέσεις των αιτήσεων. Ε, Αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν έχουν οδηγήσει σε μια κάποια μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των προγραμμάτων. Από την άλλη η χρήση των ηλεκτρονικών των μέσων αυτών είναι ελαφρώς δύσκολη και χρονοβόρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε να κάνουμε με την ενδιάμεση επανεξέταση και γι' αυτό ήδη τα γραφεία που ασχολούνται με τα προγράμματα αυτά προετοιμάζουν μια κάποια ανάλυση ε, για τα θέματα και τις πιθανότητες αλλαγών έτσι ώστε να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο το γραφειοκρατικό βάρος. Και αυτό έχει σχέση και με αυτά τα οποία είπε η κυρία Φερχέγεν και τις δυσκολίες τις οποίες ανέφερε. Θα υπάρξει λοιπόν κατά τη διάρκεια της πορείας βελτίωση της γραφειοκρατίας, όχι μόνο σχέση με την αίτηση, αλλά και τις εκθέσεις οι οποίες πρέπει τακτικά να υποβάλλονται. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Να περάσουμε τώρα στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Δρογεύσκη, ο οποίος είναι εισηγητής ε, αρμόδιος για τον προπολογισμό δύσκολο καθήκον σε στιγμές που ο υπολογισμός για το πολιτισμό και την παιδεία πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί Καλωσορίζω τη Σλοβακική Προεδρία. Γνωρίζω ότι η Σλοβακία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την παιδεία και τον πολιτισμό και σίγουρα η Προεδρία αυτή θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχω δύο ερωτήσεις όμως να σας θέσω. Καταρχάς, η Προεδρία είναι η κατεξοχήν ευκαιρία να προωθήσει κάποιο το δικό του πολιτισμό. Αυτό γίνεται είτε στις Βρυξέλλες είτε στη Σλοβακία με διάφορες ε, δραστηριότητες, καλλιτεχνικά ε, και σε εκδηλώσεις ε, και αυτό είναι εξαιρετικό. Θα ήθελα να ξέρω τι έχετε προετοιμάσει, τι σκοπεύετε να προετοιμάσετε για τη Σλοβακική Προεδρία σε θέματα πολιτισμού και να αρχίσουμε να τα διαφημίζουμε κιόλας. Ε, δεύτερο, μια πρόταση από πλευράς πολιτισμού. Το Μάρτιο, πριν από κάποια χρόνια, Είχαμε μία πυρκαγιά σε ένα κάστρο στην Κρασναχόλικα και καταστράφηκε ολοσχερός το κάστρο, αλλά και πάρα πολλά εκθέματα και χρειάστηκε να αναζητήσουμε πολύ γρήγορα τρόπο για ανοικοδόμηση αυτού του εξαίσιου αυτού ε, μνημείου. Η Σλοβακική Προεδρία σκοπεύει να αφιερώσει κονδύλια για τη διάσωση μνημείων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή καταστροφής. και αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε και σε άλλες περιοχές όταν υπήρχε για παράδειγμα σεισμό που κατέστρεψε κάποιο μνημείο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε περίπτωση που υπάρχει μια ακόμα τέτοια δραματική κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις περιπτώσεις ώστε να δράσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα. Σας έχω γνωρίσει και τους δύο όταν ε, και εγώ διατέλεσα υπουργό και ξέρω ότι θα κάνετε εξαιρετική δουλειά. Τίποτα άλλο λοιπόν. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η κυρία Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση και τις δύο παρουσιάσεις και σας ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο ε, Γκράντσα. Στην παρουσίασή σας αναφέρατε ότι μία από τις προτεραιότητές σας ε, είναι να υποστηρίξετε το ταλέντο, κύριε Πλάπτσαν. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να το επιτύχετε αυτό, δεδομένου ότι αυτοί οι ταλαντούχοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες και μάλιστα ε, ε, από πολύ νωρίς. Άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε στην ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ε, Επαγγελματικών Προσόντων και θα ήθελα να ξέρω πώς θα γίνει αυτή η αναθεώρηση ε, στη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας. Η κυρία Σβεντρόβα. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που βλέπω εδώ την ε, Σλοβακική Προεδρία. Είναι μια χώρα με την οποία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Και έχω αρκετές ερωτήσεις για σας, ε, αγαπητοί Υπουργέ, και κάποια σχόλια. Καταρχάς για τον Υπουργό Πολιτισμού. Δεν θα αναφερθώ και πάλι στην οδηγία για τα Ακουστικά μέσα, την περιγράψατε πάρα πολύ καλά και μας είπατε ακόμα και ε, εκπομπές που παρακολουθείτε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού. Ο κύριος Δρογεύσκη αναφέρθηκε και στο θέμα του πολιτισμού επίσης. Τι σκοπεύετε να παρουσιάσετε εσείς, τι νέο θα έχουμε στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτισμού. Είναι μια πρόκληση η οποία πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και πολλές εκδηλώσεις ε, θα προκύψουν και από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι βέβαιος, βέβαιη ότι το 2018 θα υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και θα μπορέσουμε να έχουμε και χρηματοδοτική στήριξη για αρκετές εκδηλώσεις ώστε πραγματικά να προσεγγίσουμε τους ευρωπαϊκούς πολίτες και να ε, προσεγγίσουμε και την ε, και διατήρηση της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς της Ευρώπης. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερο θα είμαστε προετοιμασμένοι και πρέπει να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, κατά την άποψή μου. Αυτή είναι η έκκληση, λοιπόν, που σας απευθύνω. Κύριε Πλάφτσαν, σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητές σας. Νομίζω ότι το επόμενο εξάμεινο θα αρχίσετε να ασχολείστε και με το θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Είναι πολύ φιλόδοξο σχέδιο αυτό και υπάρχει και ε, το θέμα της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης για τα επαγγελματικά προσόντα και εγγυήσει για τις νέες δεξιότητες. Αναφερόμαστε σε μία αναθεώρηση και σε κάτι εντελώ καινούριο. Δεν θα ήθελα λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, απλώς να τονίσω ότι πρόκειται για τιτάνιο έργο και το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες κατά την άποψή μου, περιλαμβάνει και μία ερώτηση, την οποία και θα σας θέσω. Το θέμα της αναγνώρισης ε, δεξιοτήτων ε, πτυχιούχων πανεπιστημίων. Ε, αγνοούμε τελείω τη διαδικασία της Μπολόνια και ελπίζω να κάνετε κάτι γιατί η διαδικασία της Μπολόνια είναι αυτή η οποία συνδέει τον πανεπιστημιακό τομέα, τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε αυτό κατά την εκπόνηση ενός νέου εγγράφου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα, θα καταρτήσουμε και σχετική έκθεση και είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις από πλευράς μας, γιατί για το μέλλον της Ευρώπης, ε, για την εκπαίδευση, για την αποσχολησιμότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ανήκω στην ομάδα των αισιοδόξων που λέγουν ότι θα είναι επιτυχής η Σλοβακική Προεδρία. Γνωρίζω και τους δύο υπουργούς και νομίζω ότι η παρουσία της είναι εγγύηση ότι αυτά τα οποία λέγουν θα γίνουν πράξεις. Θα ήθελα να εμείνω σε αυτά που είπε ο Υπουργός Πολιτισμού που ε, έθεσε το βάρος του πολιτισμού στην Ευρώπη σήμερα. Πολλές φορές στα πλαίσια των καθημερινών δυσκολιών ξεχνάμε τον πολιτισμό. Ξεχνάμε ότι η καθημερινότητά μας, ο πολιτισμός μας σε καθημερινή βάση είναι το φάρμακο για όλες τις μορφές βίαιη ριζοσπαστικοποίησης. και θα πρέπει να υπογραμμίσετε ότι το Δεκέμβριο θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Εγώ λοιπόν εμπιστεύομαι αυτά τα οποία είπατε. Για τον έτερο Υπουργό επέμεινε στα θέματα της πολιτικής για τους νέους. Εγώ ήμουνα στη συνάντηση που είχαμε οργανώσει για τους νέους γιατί δεν υπήρχε μεγάλη παρουσία βουλευτών. Είδα στο Στρασβούργο τους νέους ανθρώπους γεμάτους γνώση και επιθυμία για γνώση και ε, χαίρομαι που θα γίνει και η διάσκεψη αυτή στο Κόζιτσε, θα πάρω και εγώ μέρος και ελπίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Φίτσος στο Στρασβούργο ότι δηλαδή θέλει μια πολιτική για τους νέους και για τους πολίτες γενικά διαφανή ε, και αποτελεσματική, αυτό να είναι πραγματικότητα. Για το θέμα των ικανοτήτων, των ταλέντων, ε, ήδη έχουν τεθεί οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Με χαρά άκουσα ε, το ότι εμείνατε στην πολυπολιτισμικότητα. Το έθεσε αυτό ο κύριος Μάντεριτς. Θα ήθελα να έλθω εδώ στο θέμα των γλωσσών των μειονοτήτων. Εσείς μπορέσατε να μιλήσετε στην γλώσσα σας στο κοινοβούλιο. Εγώ είμαι Ουαλή, αλλά δεν είναι πλήρως επίσημη η γλώσσα μου εδώ και δεν είμαι σε θέση να την μιλήσω. Όταν μιλάμε λοιπόν για την καταπολέμηση του αποκλεισμού, το θέμα των μειονοτικών γλωσσών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο καθένας για να λειτουργεί ισότιμα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα. Το δεύτερο σημείο είναι ένα ευρύτερο θέμα Είπατε ότι μία από τις τρεις αρχές της Προεδρίας σας είναι τα απτά αποτελέσματα για να αποδείξουμε στους πολίτες ότι τα κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα μπορεί να βελτιώσουν την καθημερινότητά του. Όπως είπα εγώ προέρχομαι από την Ουαλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα μεγάλο τμήμα της Ουαλίας ψήφισε για να εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά το δημοψήφισμα οδήγησε σε διαφορετική κατεύθυνση. Η σχέση λοιπόν αυτή με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Σε πάρα πολλά τμήματα της χώρας μου δεν το αποδείξαμε αυτό, υπάρχουν πολλοί λόγοι ίσως γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για τον πολιτισμό και για τους νέους οι οποίοι έχουν ανάγκη να βελτιωθεί η προοπτική τους στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ερώτησή μου παραπέμπει σε μια έκθεση που συζητήσαμε σήμερα το πρωί για την προσβασιμότητα. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα δικαιώματα των ΑΜΕΑ και στην πρόσβαση και στα πολιτιστικά προϊόντα για τους τυφλούς. Επανειλημμένα, ήδη από το 2016 υπενθυμίσαμε με το ψήφισμά μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικυρώσει τη σύμβαση του Μαρακές, τη συνθήκη μάλλον του Μαρακές, για την πρόσβαση στα βιβλία των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Τρία χρόνια μετά όμως από την ψήφιση του εγγράφου αυτού έχει μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο. Ο Καναδάς είναι η τελευταία χώρα που επικύρωσε το κείμενο αυτό Νομίζω ότι είναι πραγματικά λυπηρό που σε ένα τόσο ε, σημαντικό θέμα συνένεσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συμμετέχει στη διαδικασία επικύρωσης. Είναι σουρεαλιστική η κατάσταση αυτή. Να θυμίσω ότι η Βόρεια Κορέα είναι ε, ανάμεσα στις 20 χώρες που έχουν ε, επικυρώσει την σύμβαση αυτή. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Η πρώτη, η Προεδρία σας θα προσπαθήσει να ξεμπλοκαριστεί το εμπόδιο αυτό έτσι ώστε να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν τη συγκεκριμένη συνθήκη. Και θα ήθελα να μάθω επίσης ε, αν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των ρυθμίσεων για την πνευματική διοκτησία ε, θα αναλάβετε την υποχρέωση έτσι ώστε οι προβλέψεις της συνθήκης του Μάρακες να συμπεριληφθούν στην νέα νομοθεσία. Και τελευταίος ο μιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρουσιάσατε τις προτεραιότητές σας και προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερους που ανάμεσα σε αυτές τις προτεραιότητές σας συγκαταλέγεται και αθλητισμός. Και ή προτεραιότητε και διπλωματία ε, για τον αθλητισμό και σε ό,τι αφορά και το θέμα των ε, προσφύγων. Χαίρομαι ιδιαίτερω επίση, για το γεγονός ότι μιλάτε για την εξέβρεση ταλέντων και για την προώθηση και προαγωγή του ταλέντου στην κοινωνία μας. θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, την κατάρτιση τέτοιων ατόμων και όχι μόνο στον τομέα του αθλητισμού αλλά και σε άλλους τομείς. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά αυτή την διτή εκπαίδευση. Τι εμπειρίες έχετε να μας παρουσιάσετε και ποια προσέγγιση θα ακολουθήσετε σε ό,τι αφορά την πρόθεση ταλέντου και την εξάφρυση ταλέντου μεταξύ των ένων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Θα δώσω το λόγο στους υπουργούς πάλι να προσθέσω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς είδατε με πόσο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την παρουσίασή σας. Είδατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και γι' αυτό θα ήθελα να μπορούμε να υπολογίζουμε στη Σλοβακική Προεδρία στα τρία μεγάλα θέματα, κυρίως την οδηγία VMS Το Σεπτέμβριο θα γίνει η πρόταση από πλευράς της Επιτροπής μας. Θα εργαστούμε στον ενδιάμεσο χρόνο ε, έτσι ώστε πριν από το τέλος του ενεστώτος έτους να κλείσουμε κάτω και από τη δική σας Προεδρία την θέση του Κοινοβουλίου και ζητάμε την υποστήριξή σας ιδιαίτερα για τα θέματα τα οποία έχουμε αναφέρει, το λεγόμενο level playing field όπως επίσης και για το θέμα της ρητορικής μίσους. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ενισχυθούν στο πλαίσιο της VDMS και όχι να αφαιρεθούν. Υπάρχουν και άλλα θέματα πάνω στα οποία έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να έχουμε μια κάποια συμφωνία. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Έτος, και θα δώσω εδώ το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την πολιτιστική κληρονομιά για το 2018. Η πρόταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθυστερεί. Περιμένουμε την πρόταση από πλευράς της. Γνωρίζουμε ότι οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι προβλέψεις αυτές να ολοκληρωθούν εγκαίρως και δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ στον προϋπολογισμό του 17. Συνεπώς λοιπόν ε, και σε συνεργασία με τον συνάδελφο σας ζητάμε να μας βοηθήσετε. Δεν είναι δυνατόν μετά από τη σκληρή μάχη που δώσαμε έτσι ώστε το 2018 να κηρυχθεί σαν σημαντικός χρόνος για τον πολιτισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στην ανθρωπότητα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχουν προβλέψει έστω και ένα ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο μειώνουμε τα προγράμματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας που είναι ανεπαρκή ε, και τα κάνουμε ακόμα λιγότερο ε, αποδοτικά. Τρίτη ερώτηση είναι το θέμα της πολιτιστικής διπλωματίας. Θα πρέπει να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα εμένει ιδιαιτέρως. και θέλουμε εμείς να καταθέσουμε και μία πρόταση πιλωτική για την κρίση και την καταστροφή της, ε, πολιτισ... Ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Μεσογειακή Λεκάνη. Νομίζω ότι Είχαμε επίσης ε, και μία συνάντηση με την διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με τις χώρες μας ΦΕΚ. Ήδη συναντηθήκαμε και με αρχαιολόγους Σύρους, ένας από αυτούς είναι εξόριστος στο Στρασβούργο. Συναντηθήκαμε επίσης και με εκπροσώπους α, ε, ε, τρισδιάστατων εικόνων και ε, αεροσκαφών φωτογραφικών χωρίς πλήρωμα, τα οποία ελέγχουν αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Παλμύρα μετά τις επιθέσεις, διότι δυστυχώς υπάρχει αυτό που θα λέγαμε πλιάτσικο ουσιαστικά των αρχαιοτήτων, ακόμα και από τους στρατιωτικούς του καθεστώτος Ασάντ. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα και να καλύψουμε το κατεπήγον θέμα, έτσι ώστε η πιθανή ανοικοδόμηση κάποιων πολιτιστικών αγαθών να μην συνεχιστεί. Ε, και θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει το ταχύτερο δυνατόν και την οδηγία για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών στην Ευρώπη από τρίτες χώρες. Την περιμένουμε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Τέλος, ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο αθλητισμός. Εμείς ε, έχουμε προχωρήσει με μια έκθεση, έχουμε επίσης κάνει και μια προετοιμασία για το θέμα της διπλής σταδιοδρομίας. Υπάρχει επίσης κάτι το επίγον το οποίο πρέπει να σας το μεταφέρουμε και αφορά στον προϋπολογισμό. Το Εράσμος κυρίως πρέπει να προστατευθεί. Έχουμε πετύχει κάπως περισσότερα χρήματα. Αλλά το Creative Europe και η Ευρώπη για τους πολίτες είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσει οι οποίες υπάρχουν. 11% μόνο των προγραμμάτων που έχουν κατατεθεί θα χρηματοδοτηθούν από ό,τι φαίνεται. Το 17 για την Ευρώπη των πολιτών πρέπει να αλλάξουμε την τάση αυτή, είναι απαράδεκτη. Θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο εκθέσεις εφαρμογής όλων αυτών των προγραμμάτων. Θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε και ελπίζω έτσι να βοηθήσουμε και την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσανατολίσουν καλύτερα την ενδιάμεση αξιολόγησή τους το 2018. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν, νομίζω ότι έπρεπε να σας τα θυμίσω αυτά. Υπάρχει εν πάση περιπτώσει μια κοινή στρατηγική την οποία πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Πρώτα ο κύριος ε, Μάνταριτς και μετά ο κύριος Πλάβτσαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε ευχαριστώ και για τις ενδιαφέρουσες αυτές ερωτήσεις και προτάσεις που μας κάνατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον, την φίλη μας, την ε, ε, κυρία Ευρωβουλευτή Μόλικοβα, για την υποστήριξη που εξέφρασε. Ελπίζω ότι και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της Σλοβακικής κυβέρνησης θα σας απογοητεύσουμε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους όσους έχουν υψηλές προσδοκίες σε ό,τι αφορά τη Σλοβακική Προεδρία ο κ. Μπογκάν και το ερώτημα που έθεσε για την, το θέμα του πολιτισμού στην Μέση Ανατολή ιδιαίτερως και είχα συνεργαστεί μαζί σας, αποτελέσατε μοντέλο για εμένα σε ό,τι αφορά και την αναζήτηση ε, πόρων για τον πολιτισμό. Το θέμα των πολιτισμικών εκδηλώσεων τώρα. Αμφίβολα, μια και μιλάμε για το θέμα τη πολιτισμική διπλωματία εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για, την... Ε, για τι υπόλοιπε χώρε, ο πολιτισμό αποτελεί ένα θέμα ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μια μικρή χώρα, ιδιαίτερα όπω η Σλοβακία, που είναι σε μεγάλο βαθμό και αφανή κάπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μεγάλο μεγάλο όγκο εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Σλοβακία και ίσως να προσέξετε και ότι διοργανώθηκε και μια συνευλία στις 7 Ιουλίου στις Βρυξέλλες στην έναρξη της Προεδρίας. Είναι καλή συνεργασία με την ε, Ολλανδική Προεδρία πριν από κάποιες εβδομάδες σε ένα σύγχρονο μουσείο στην ε, Σλοβακία, στην Πρατισλάβα, ξεκίνησε ε, μία κοινή έκθεση ε, με την οργάνωση Κόμπρα. Από κοινού με τις κάτω χώρες συμμετείχε μάλιστα και η πριγκίπισσα των κάτω χωρών. Και έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα που έθεσε η Προεδρία των Κατοχωρών προκειμένου να ευωδώσουν τώρα κάποιες ε, προσπάθειες νομοθεσίας μεταξύ άλλων και οι νομοθεσίες που αναφέρεται. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με, τις, ε, με την Τρόικα, με τις ε, χώρες της Ολλανδίας και της Μάλτας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα κάνω και τα εγγένεια μιας μεγάλης γοθικής έκθεσης από πλευρά ε, της ε, Σλοβακίας. Δεν θέλω να σας ε, κουράσω με λεπτομέρειες, αλλά έχουμε ζήσει και διάφορες καταστροφές ό,τι αφορά εκδηλώσεις πολιτισμικές. Γι' αυτό λοιπόν να εκτιμούμε την υποστήριξη και από, άλλων, από άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τα έργα τέχνης τα οποία έχουν καταστραφεί. Η κυρία Σόντροβα έθεσε το ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς το 2018. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα αναμένουμε την ακριβή διατύπωση της πρότασης την οποία θα υποβάλει ο Επιτροπός και μόνο τότε θα ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα, το οποίο προς την παρούσα φάση δεν έχει ακόμα σαφήνεια. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κυρίω. αν δεν έχουμε επαρκή πόρους, θα είναι διακοσμητικό μόνο αυτό, καταλαβαίνετε, ως τίτλος. Εμείς αποκινούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιθέμεθα να συνεργαστούμε προκειμένου να δούμε τι θα γίνει αν αυτό θα σημαίνει μεταφορά κεφαλαίων και πόρων μεταξύ των ε, γραμμών του προπολογισμού. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω στην παρούσα φάση, αλλά αυτή τη στιγμή θα έχουμε θέσει όλε τι προτεραιότητε επιτάπητο. Θα χρειαστούμε τη σωστή χρηματοδότηση. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα θέματα που συνδέονται με το έτος πολιτισμικής κληρονομιάς ε, δεν περιορίζονται ε, στα θέματα πολιτισμού και των εκδηλώσεων. Τίθενται και οικονομικά θέματα, δημοκρατικά θέματα, ε, οικονομικά ζητήματα και όλο το ευρύτερο πλαίσιο και συγκείμενο της κοινωνίας μας. Θίξετε τώρα το θέμα των μηνωτικών γλωσσών, το οποίο αφορά και πολλές χώρες με μεγάλους πληθυσμούς μειονοτικούς με τα δικαιώματά τους ασφαλώς ό,τι αφορά τη γλώσσα τους, ό,τι αφορά τον πολιτισμό τους. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Προεδρίας δεν πρόκειται να γνωρίσουμε και να αφήσουμε κατά μέρο το ζήτημα αυτό. Στη Σλοβακία δεν προετοιμάζουμε στην παρούσα φάση ένα ειδικό πολιτισμικό ταμείο για την προώθηση των πολιτισμών των μειονοτήτων. Σε αυτό αυτό το πρόγραμμα συγκαταλέγεται και η προώθηση των γλωσσών των μειονοτήτων. Και θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι ιστορικός πώς είναι η πρώτη φορά που στη Σλοβακία έχουμε συμμαχία α, μεταξύ Σλοβακικής, Σλοβακικού κόμματος και Μηνωτικού Ουγγρικού κόμματος. Η κατάσταση λοιπόν είναι αρκετά θετική από αυτή την άποψη. Ο κύριος Ζούλο έθεσε το θέμα της προσβασιμότητας και της ε, συμφωνίας του Μαρακές. Και εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα της πτυχής των ατόμων με αναπηρία. Και ξέρουμε ότι το θέμα αυτό προς το παρόν είναι μπλοκαρισμένο, αλλά μετά από την απόφαση που θα λάβει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ακόμα εκκρεμεί η απόφαση αυτή, τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα χαρούμε να συζητήσουμε την πρόταση της Επιτροπής και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις προκειμένου η συμφωνία να επικυρωθεί το σύντομα δυνατό. Ελπίζω έτσι να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Υπουργός Πλάβτσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα του ταλέντου. Κύριε Πέντα, κυρία Σμόλκοβα, κύριε Λιπάτσκα, με ρωτήσατε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η ανισότητα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και γνωρίζουμε ότι οι ανισότητες ε, αργότερα έχουν αρνητικές συνέπειες ε, για ε, το σύνολο της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό ακριβώ η Σλοβακική Προεδρία έχει θέσει ένα, ως ένα από τα κύρια θέματα τους το ταλέντο, την ανακάλυψη του ταλέντου και από εκεί και πέρα όχι μόνο την ανάπτυξή του σε άτομα τα οποία επιδεικνύουν ταλέντο στον αθλητισμό ή στα μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο, μαθητές που ήδη συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ε, διεθνούς ε, εμβέλειας. Θέλουμε να ανακαλύψουμε ταλέντο, ε, το ατομικό ταλέντο του καθενός. Να βρούμε και να επιλέξουμε κάτι μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός ατόμου και να βρούμε τρόπους να το αναπτύξουμε αυτό το ταλέντο και να, δείξουμε, να αναδείξουμε τη μοναδικότητα του καθενός και να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν σε κάτι συγκεκριμένο στη συνέχεια της ζωής τους, σε κάτι εξαιρετικό. Θα υπάρξει και σχετική διάσκεψη για το θέμα για την ανάπτυξη και υποβοήθηση του ταλέντο ε, το Σεπτέμβριο στην Κόζιτσα και εκεί θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε ότι σε αυτό το φόρουμ, όπου θα υπάρχει και μεγάλη εκπροσώπηση εμπειρογνωμόνων, θα συζητηθούν ευρύτατα τα θέματα αυτά. Το ταλέντο αυτών που έχουν ήδη επιδείξει ότι υπάρχει κάποιο ταλέντο, αλλά και πώς μπορούμε να αναδείξουμε ένα ταλέντο που δεν έχουμε ανακαλύψει ίσως τα υπόλοιπα παιδιά για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια τη ζωή τους. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, για τις δεξιότητες, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η κατάσταση στην αγορά εργασία εργασίας ε, απαιτεί συνεχώς νέες δεξιότητες. Οι εργοδότες δεδομένης και της πρόοδου απαιτούν ε, συνεχώς από τους εργαζομένους τους ε, διαφορετικές και νέες δεξιότητες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο μαζί με το εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόοδος και να μπορέσουμε να συγκρίνουμε δεξιότητες και να διευκολύνουμε την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που είναι και ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βοηθήσουμε την βελτίωση και την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων ώστε να αποτελέσει καλύτερο γνώμονα. Γι' αυτό και ακριβώ ε, και εμεί, ως Σλοβακική Προεδρία θα μεσολαβήσουμε ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία όταν θα συζητηθεί η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων. Όσον αφορά τι ερωτήσει της κυρίας ε, Σμόλκοβα, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του θεματολογίου ε, και της δέσμης Μέτρους για τη δεξιότητε, θα παρουσιάσει του χρόνου ένα σχέδιο εξυγχρονισμού της διαδικασίας εκπαίδευσης και ίσως και βελτίωση της διαδικασίας της Μπολόνιας. Ε, εγώ εκπροσωπούσα τη Σλοβακία στην ομάδα παρακολούθησης ε, της ε, Μπολόνιας ευθύ εξ αρχής και έχουμε παρακολούθησει πολύ αναλυτικά τα συμπεράσματα αυτής της ομάδας, η οποία συναντάται δύο φορές το χρόνο και θα συζητήσουμε και κάποιες επικαλύψεις, ίσως και το σχετικό έγγραφο της ευρωπαϊκή Επιτροπής για τον εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη διαδικασία της Μπολόνιας. Προσπαθούμε να βρούμε επαφές, διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει σχετικά έγγραφα. Ε, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα στον τομέα του εξυγχρονισμού, βελτίωση της ε, ποιότητας των διδασκόντων, της ίδιας της παιδείας, εμείς ως Προεδρία θα εξετάσουμε τις συνέπειες ε, των πανεπιστημίων και της ανώτατης εκπαίδευσης ε, στις περιφέρειες, προσπαθώντας να βρούμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ περιφερειών και επιχειρήσεων ή και κρατικών τοπικών αρχών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες συνέργειες για την ανάπτυξη των περιφερειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις διευκρινήσεις και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα, επειδή αρκετοί συνάδελφοι και υπήρχε και σχετική έκκληση και από τους υπουργού και από την υποφαινομένη. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να σχολιάσει τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Ξέρω ότι έχουμε τον κύριο Φίλιπ Βαντεπούλ εδώ, τμήματάρχη της ΕΑΚ. Αν μπορείτε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας μετά από τη συζήτηση που προηγήθηκε. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε επανειλημμένα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2018. Έχουμε προχωρήσει στην επεξεργασία της πρότασης Ελπίζω να μπορέσετε να την δεχτείτε σε έφετο χρόνο, έτσι ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από το Σεπτέμβριο υπό τη Σλοβακική Προεδρία να ξεκινήσουν τη δουλειά. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις σας συστηματικά. Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν γρήγορα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις οι οποίες ε, θα πρέπει να ληφθούν, να ληφθούν γρήγορα για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα την 1η Ιανουαρίου του 2018. Ένα πράγμα να προσθέσω, ε, το θέμα του προϋπολογισμού. Ξέρω ότι υπάρχει μια ε, αιμονή από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για την, για το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε ακόμα λίγους μήνες για να βρούμε μια λύση για κατάλληλη χρηματική κάλυψη. Κοιτάξτε, πρέπει να επιμείνουμε πολύ για να κερδίσουμε στον τομέα του πολιτισμού. Πάντως θα ήθελα να είναι ευαίσθητη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρά πιο γρήγορα. Πριν δώσω το λόγο στην Κάμερα Εβέρτ να πω ότι είναι μια νομοθετική διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρος και εγώ πιστεύω ότι θα μας κάνετε την πρότασή σας πριν από τον μήνα Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γραμμέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ να παραδεχτώ ότι μπήκα σε πειρασμό να πάρω το λόγο. Μα δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο δύσκολο, αν ξέρουμε ότι όλοι συμφωνούν. Το Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο ε, συμφωνούν. Και τις παίρνει τη Επιτροπή Μήνε. και μετά μας λένε «Α, τώρα βιαστείτε όμως» και ασκείται πίεση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και για να βιαστούμε. Ε, πιστεύω ότι είναι κάπως... Ε, ακατάλληλη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μήνε για να καταθέσει την πρόταση και εμεί τελευταία στιγμή πασχίζουμε να τρέξουμε τελευταία και καταϊδρωμένη. Και το Συμβούλιο δηλαδή. Μόνο και μόνο επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να υποβάλει α, στο σωστό χρονικό διάστημα, γρήγορα, μία σχετικά απλή πρόταση. Και κοιτάξτε, το 2018 δεν είναι τόσο μακριά. Μα και τα κρατη δεν χρειάζονται χρόνο να προετοιμαστούν. Δεν πρέπει και αυτά να προβλέψουν τους πόρου στους προπολογισμού τους. Παρακαλώ λοιπόν, κατεπηγόντω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα να μας υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την πρόταση αυτή. Να ξεκινήσουμε επιτέλου τις εργασίες μα. Νομίζω ότι αυτό βρίσκει τους πάντες σύμφωνους ε, και το Συμβούλιο από αυτά που ακούσαμε και από τον Υπουργό και επίση θεωρώ ε, ότι επειδή για το Ευρωπαϊκό έτος του 2018 αναφερθήκαμε ε, και στο παρελθόν, μετά σταμάτησαν οι συζητήσεις, μετά τα ξανά ξεκινήσαμε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια εξαιρετική ομάδα όλων των κυβερνήσεων και έχει γίνει το προπαρασκευαστικό έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε και τις προτάσεις εγκαίρως. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε έναν τρόπο να επιταχύνουμε και εμείς τις δικές μας εργασίες, αλλά ελπίζαμε να έχουμε τις προτάσεις μέχρι τον Ιούλιο. Και είναι και σοβαρό αυτό, διότι ε, επιτέλους καταφέραμε να έχουμε αυτό το έτος και με την υποστήριξη του Πρόεδρου Σούλτς, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλεγε τίποτα επί του ζητήματος και θα ήθελα ε, να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο, χωρίς να θέλω να επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι για το 2017, αλλά γιατί μας ενδιαφέρει και το 2018. Τα διάφορα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται, θέλουν να συνεργαστούν, θέλουν να προωθήσουν και κάποιες προτάσεις. Επομένως, πραγματικά σας ζητώ να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αυτά, αλλά γιατί νομίζω ότι έγινε αντιληπτή. Τώρα, αν χρειαστεί θα αποστείλω και επιστολή στον Επίτροπο, διότι νομίζω ότι πλέον ε, τα πράγματα να γίνουν ε, όπως πρέπει και δεν θα θέλαμε να φτάσουμε τέλη Σεπτεμβρίου και να μην υπάρχει πρόταση. Αποκλείεται αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν να το διαβιβάσετε και στον Επίτροπο αυτό. Ολοκληρώνουμε με αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, τη διάθεσή σας, ε, αγαπητοί Υπουργοί. Όπως θα βλέπετε εδώ υπάρχουν προτάσεις, σαφείς ιδέες, ε, ε, ζωηράδα και θέλουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Και ελπίζω και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως να προσδώσουμε τη δέουσα προσοχή στα θέματα αυτά και να προωθήσουμε αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. we have a very important thing to... Συνάδελφοι, έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ακόμα. Διότι τώρα έχουμε την έκθεση για τον προϋπολογισμό, σχέδιο έκθεσης για τον προϋπολογισμό. Παρακαλώ. Five minutes. Two minutes. Two minutes. Δύο λεπτά Λοιπόν, έχουμε τώρα το πολύ σημαντικό προσχέδιο που υπέβαλε ο εισηγητής αρμόδιος για τον προπολογισμό του 2017, ο κ. Ντρογεύσκη. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία προβλέπει τρεις γνωμοδοτήσεις ε, γνωμοδότηση για την εντολή για τον τριμερή διάλογο, την οποία εγκρίναμε ήδη τον Ιούνιο. Αυτή είναι η γνωμοδότηση για το πρώτο ψήφισμα που δίνει εντολή για διαπραγμάτευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων για τη διαπραγμάτευση και το επόμενο βήμα, το τελευταίο, θα δοθεί το Σεπτέμβριο, όταν θα ψηφίσουμε επί των τροπολογιών. Προθεσμία για τις τροπολογίες 14 Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Το ξέρω ότι πιέζει λίγο η διορία, αλλά το είχαμε ε, πει σε όλους τους συναδέλφους ήδη ε, από την 1η Ιουλίου. Το είχαν αποφασίσει οι συντονιστέ και το διαβιβάσαμε σε όλου την 1η Ιουλίου. Παρακαλώ να σεβαστείτε την προθεσμία. Αλλιώ, εάν δεν προλάβετε, μπορείτε να υποβάλλετε επισήμω ε, ε τροπολογίε στην Επιτροπή Προπολογισμών μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, δεν κάνω λάθο. Τώρα. Επαναλαμβάνω προθεσμία αύριο 2 η ώρα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σδρογεύσκη αμέσως και κατόπιν στους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Στρογεύσκη. Pani Przewodnicząca, szanowne koleżanki. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην ε, διάθεσή μας, έχει πάει 11 και 25. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι και σύντομο. Θα επικεντρωθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία της έκθεσης. Α. κοιτάξουμε λοιπόν καταρχάς τις διαδικασίες. Ε, η κυρία Πρόεδρο, ήδη σα ενημέρωσε σε ό,τι αφορά τις ε, προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών. Είναι πραγματικά απλισμένα τα πράγματα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και να έχουμε επίση υπόψη ότι η κατάρτιση της γνωμοδότησης συνοδεύτηκε και από μεγάλη πίεση. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Και αυτό ισχύει για πολλούς εισηγητές, οι οποίοι έπρεπε να καταρτήσουν την γνωμοδότηση παρά το γεγονό ότι δεν είχαμε ακόμα το σχέδιο προπολογισμού. Εγώ δεν περίμενα τη δημοσίευση του σχεδίου του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβάστηκε τα τι προθεσμίε, αλλά τελευταία στιγμή τα κατέθεσε όλα και η γνωμοδότηση είχε προετοιμαστεί βάσει όμως του σχεδίου του προπολογισμού και όχι βάσει των προσδοκιών. Και πρέπει να σας πω ότι με ικανοποιεί το ποσό που προβλέπετε για το Erasmus Plus. Δεν έγιναν περικοπές, και μάλιστα έγινε 16% αύξηση, η πιο υψηλή αύξηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Erasmus Plus, οι εκκρεμείς ε, δεσμεύσεις περιορίστηκαν και ε, μειώθηκε η ιστεροβαρής ε, χρηματοδότηση και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δεν είναι τα πράγματα, ξέρετε, τόσο ρόδινα σε όλους τους τομείς. στη Europe for Citizens ε, έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση. Αλλά επειδή δημιουργήθηκαν αποθεματικά για άλλα προγράμματα, οι αλλαγέ αυτέ δεν μα ικανοποιούν πλήρω. Και χθε μίλησα με την κυρία Φώστερ. Φώστερ, συγγνώμη. Και συμφωνήσαμε για μια συγκεκριμένη στρατηγική. Το ποσό λοιπόν, το εν λόγω ποσό, είναι μάλλον μικρό, ωστόσο είναι κρίσιμο για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, να παρατηρήσουμε ότι κάποια στοιχεία λείπουν λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για κάποια πολιτικά προγράμματα. Κάποια πολιτικά προγράμματα στεφτήκαν με επιτυχία. Δεν είναι δυνατόν όμω να υπάρξει μόνιμη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν πόροι προ την κατεύθυνση αυτή. Και επιπλέον δεν λάβαμε νέου πόρου για νέε προπαρασκευαστικέ δράσει και για πολιτικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε τα εξή. Η παρουσίαση του σχεδίου προπολογισμού καθυστέρησε. Και αυτό ισχύει και για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Και το Κοινοβούλιο έχει θέσει κάποιε προθεσμίε οι οποίε είναι πραγματικά ε, δεν μα επιτρέπουν να δουλέψουμε σωστά. Δουλεύουμε υπό πίεση με έναν πραγματικά ρυθμό απάνθρωπο. Κατά δεύτερον, καλωσορίζουμε τι αλλαγέ σε ό,τι αφορά το Erasmus Plus. Δεν είναι τεράστια επιτυχία, παρ' όλα αυτά είναι επιτυχία. Είναι ένα επίτευγμα αυτό. Κατά τρίτον, εκφράζουμε ανησυχία. Ανησυχία γιατί δεν προβλέπεται περιθώριο για τα πιλωτικά project, για περαιτέρω ενίσχυση των πόρων που χρηματοδοτούν τα πιλωτικά προγράμματα. Και αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία και την ε, μεταναστευτική κρίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε σαφώς το ρόλο της πολιτισμικής διπλωματίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή της στην ανάγκη αυτή και αυτό το καλωσορίζουμε. Τέλος, όπως είπε και η κυρία Κάνβελτ, αυτό που χρειάζεται κατεπηγόντως είναι πόροι για το 2018. Και αυτό γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος πολιτισμικής κληρονομιάς. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτά. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Υπογραμμίσατε κάποια σημεία σχετικά με τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε για τον προϋπολογισμό του 17. Θα το συζητήσουμε το θέμα και με τους συντονιστές γιατί έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα στον τίτλο 3 κάποιες απαράδεκτες καταστάσεις, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και επαναλαμβάνω τα προγράμματα Creative Europe και η Ευρώπη των πολιτών είναι υποχρηματοδοτούμενα και αυτό προκαλεί μια τεράστια δυσθυμία από πλευράς των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ανεβάσουμε το όριο γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Θα προκαλέσουμε έναν πόλεμο ανάμεσα στους φτωχούς ουσιαστικά. Θα δώσω τους, στους κοιόδης το λόγο ο κύριος Μόργαν ο πρώτος. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια περίοδο θα έλεγα πολύ περίπλοκη και αυτό φαίνεται και από το Brexit. Ζητάμε πάντα όμως από τον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και του πολιτισμού κάποιες λύσεις. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τις δυνατότητες στους τομείς αυτούς να ανταποκριθούν. Απαιτείται λοιπόν σωστότερη και καταλληλότερη χρηματοζώτηση. Ε, συμφωνώ με αυτά τα οποία υπόθεσαν, για το Erasmus Plus και την αύξηση. Αλλά με το Creative Europe και την Ευρώπη των πολιτών έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα πρέπει λοιπόν να ακουστούν αυτά τα οποία λέγουμε. Αν για τους τομείς αυτούς έχουμε συγκεκριμένους στόχους, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πόροι για να πετύχουμε τις προτεραιότητες αυτές είναι ανεπαρκείς προφανώς. Πρέπει να τεθεί το ερώτημα λοιπόν, γιατί αλλιώς έχω την εντύπωση ότι το θέμα νομίζουμε ότι θα διορθωθεί μόνο του, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί βέβαια, Νομίζω λοιπόν ότι η πλειοψηφία των μελών εδώ συμφωνεί με τα μέτρα για μια σωστή απασχόληση των νέων, ποιοτική απασχόληση των νέων που θα συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της οικονομίας και μέσα από τον πολιτισμό. Συνειδητοποιούμε επίσης ότι αν πράγματι θέλουμε οι νέοι σήμερα να έρθουν κοντά στην Ευρώπη, να συμμετέχουν στα κοινά, και να προωθήσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, το θέμα του πολιτισμού είναι, θα έλεγα, κάτι που επιβάλλεται από μόνο του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε με διαφορετικό μάτι ε, και ε, το, αθλητικά, τις αθλητικές δραστηριότητες, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη σχέση αυτών των δραστηριοτήτων με τους πρόσφυγες Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να γίνουν προτάσεις και να πετύχουμε αποτελέσματα. Αυτό είναι η πραγματική δημιουργική Ευρώπη και η Ευρώπη των πολιτών. Ε, κάτι για το Erasmus Plus. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με κάποιες εθνικές υπηρεσίες, γιατί στο Βέλγιο, σαν παράδειγμα, φτάνουν και τα αιτήματα των ΜΚΙΟ. Ε, το πρόβλημα δεν είναι ένα βελγικό πρόβλημα, είναι ένα γενικότερο θέμα και γι' αυτό ίσως ένα κομμάτι ε, του προϋπολογισμού να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο για να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ειδικά στο Βέλγιο. Για την πολιτιστική διπλωματία όλοι το αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντική. Όμως βλέπουμε ότι ε, το Ευρωπαϊκό Έτος για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία η οποία θα είναι απαραίτητη, ακόμα όμως δεν έχουμε στοιχεία. Τώρα για τα προπαρασκευαστικά και πιλωτικά προγράμματα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις αξιολόγησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιβάλλουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα με την Επιτροπή. Ε, δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε περισσότερο για να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια κάποια λύση. Να προσθέσω εδώ ότι τα θέματα προϋπολογισμών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών είναι σε μια φάση ευαίσθητη. Πρέπει όμως να δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε, γιατί μερικές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι στην ουσία περιοριζόμεθα σε μια κάποια κριτική και πέραν τούτου δεν, όχι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό, πρέπει να δούμε τα αρνητικά σημεία, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έτσι ώστε τα κρίσιμα αυτά σημεία να ξεπεραστούν. Λοιπόν, κύκλος ε, είναι φαύλος διότι φοβάμαι ότι και του χρόνου και το 18 και το 19 τα ίδια θα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριος ε, Δραμπόσκι, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να προφέρετε το επιθετό μου. Έχω συνηθίσει να το λένε λάθος. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σδρογεύσκη, ο προπολογισμό θα πρέπει να συζητάτε διεξοδικά σε κάθε κοινοβούλιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συζητήσει αυτές περνάνε παρατήρητε και ε, γίνονται για του τύπου. Υπάρχει μια πραγματική συζήτηση που διεξάγεται στο Συμβούλιο. Εκεί κάθε χώρα προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντά της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει συνέχεια αυξήσει του προπολογισμού. Και η Βουλγαρία θα ήθελε αύξηση του προπολογισμού για τη χώρα μου, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές και να κρίνουμε πού μπορούμε και πρέπει να δαπανούμε περισσότερα και πού δεν θα έπρεπε να δαπανούμε περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η μηνιαία μεταφορά μεταξύ Βρυξέλλες και Στρασβούργου είναι μια πολύ δαπανηρή πολιτική λύση. Πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να δούμε πού μπορούμε να έχουμε αύξηση κονδυλίων και πού δεν μπορούμε να έχουμε. Η πολιτική μου ομάδα ζητά βιώσιμη χρηματοδότηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάλληλοι ε, σπόρους από μεγάλα, ε, για μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Για μένα οι περισσότερες προκλήσεις, ιδιαίτερα και εν ώψη του Brexit, είναι άλλε. Οποιαδήποτε επένδυση σε παιδεία, κατάρτιση, έρευνα μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση θέσεων εργασία. Δεν είναι απαραίτητο να αυξήσουμε ε, μηχανικά τον προπολογισμό. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε προγράμματα και έργα τα οποία θα μας ε, δώσουν και κάποιο αντάλλαγμα για την επένδυσή μας. Ευχαριστώ η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των τριών μεγάλων προγραμμάτων μας. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις από αυτόν και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ε, αύξηση στον προπολογισμό του Erasmus ε, ΣΥΝ, δεν νομίζω ότι αρκεί, διότι είδαμε ότι για το προσφυγικό ζήτημα και δικαίως το Erasmus Plus και το Creative Europe ε, Europe ε, έχουν νέες προσκλήσεις για να ε, εργαστούν ε, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης αυτών των προγραμμάτων. Επομένως προτείνουμε αύξηση του προπολογισμού του Erasmus 5 κατά 15% και της Δημιουργικής Ευρώπης Επίτης και να τα βελτιώσουμε αυτά γιατί υπήρχε περικοπή του προπολογισμού κατά 20%. Ακόμα και αν πάμε πάνω από τα ανώτατα όρια, εμείς επειδή ως Επιτροπή Επιτροπή Πολιτισμού δεσμευόμαστε ε, και βάσει του επιχειρήματο ότι θα πρέπει να ζητούμε προπολογισμό υψηλότερο για αυτά τα προγράμματα, πρέπει να το κάνουμε. Κατόπιν, προτείνονται αρκετά πράγματα για πιλωτικά προγράμματα, αλλά θα ήθελα να προσθέσω διότι προφανώς ε, και θα υπάρξει και κοινό πιλωτικό πρόγραμμα και σχετική πρόταση για τις εργασίες του Euronet και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκρινίσουμε ότι εμείς ζητούμε και πιέζουμε να υλοποιηθεί αυτό και ε, δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε εκτέλεση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μην λαμβάνει υπόψη τη στο Euronet. Χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και αυτό το δίκτυο ραδιοφώνου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, χρειαζόμαστε πάρα πολύ σαφή δέσμευση από την Επιτροπή Προελιτισμού προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βεβαίω και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι στον προπολογισμό αυτό. Ο κύριο Μαραγκάλ. Sí, Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πολύ τους καταρχάς με αυτά που έλεγε η κυρία Τρούπελ για τις συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά θέλουμε και κάτι πιο γενικό εδώ. Εδώ, σε αυτόν τον προπολογισμό, εργαζόμαστε λίγο στο κενό. Δεν έχουμε πρόταση του Συμβουλίου ακόμα και απλώς υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο τελικό αποτέλεσμα, κάπως θετικό, αλλά με πάρα πολλές αβεβαιότητες. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα τις λύσουμε. Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι είμαστε στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και επομένως το απόλυτο όριο που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την αναθεώρηση ε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές μας, όπως οι δικοί μας, θα πρέπει ε, να το εκμεταλλευτούν και να ε, εκφράσουν τη μεγαλύτερη φιλοδοξία, γιατί είμαστε στη διαδικασία της αναθεώρησης και πρέπει να φτάσουμε μέχρι το μέγιστο όριο που μας επιτρέπεται από νομική σκοπιά και λόγω και των οικονομικών πιέσεων, που είναι και οι πιο πιεστικές. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η γνωμοδότηση που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι θετική, μπορούμε να την υποστηρίξουμε και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πρόταση αύξησης κατά 16% για το Erasmus ε, Plus συνάδει απόλυτα με αυτό το οποίο προβλεπόταν. Δεν είναι καμιά καινοτομία. να μην είμαστε και τόσο πια ευτυχείς, γιατί αυτή τη δέσμευση είχαν αναλάβει. Και συμφωνώ και με την κυρία Τρούπελ ότι πρέπει να υπάρχουν συνέργειες το Erasmus, το European Social Forum, το Creative Initiative, όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν γιατί εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις στρατηγικές μας και τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει ε, να έχουν τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιήσουν καλύτερα αυτούς τους πόρους. Είναι πολλά τα χρήματα και δεν ε, απορροφούνται πάντα πολύ καλά για να απαντήσουν στα προβλήματα ανεργίας και την κοινωνική κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαραγκάλ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΑΚ, Φρεντερίκ Φιμάιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημής σημειώνει τα διάφορα σημεία τα οποία προτάθηκαν και την πρόταση του κειμένου και θα θέλαμε να σας επενθυμίσουμε ότι όντως ε, ο προπολογισμό για το Erasmus Plus θα αυξηθεί σημαντικά και διαπιστώνεται για το 2017 αυτή την ε, αύξηση την οποία πραγματικά περιμένανε οι διάφοροι stakeholders και οι δικαιούχοι. Αυτό θα συνεχίσει μέχρι το 2020 και τελικά ε, πετύχαμε λοιπόν αυτή την αύξηση και μάλιστα στο επίπεδο το οποίο προβλεπόταν στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση. Για, τα... για τις πληρωμές, ε, για τις πληρωμών σε ό,τι αφορά το backloading, ε, η κατάσταση πλέον σταθεροποιείται, άρα το 2017 λίγο πολύ θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δεσμέσεις πληρωμών και σε ό,τι αφορά τα, το Erasmus Plus και το Creative Europe. κατά πόσον έχουν πρόθεση και υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουμε το ανώτατο όριο για τον τίτλο 3. Αυτό ε, διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αλλιώς εμείς δεν θα έχουμε περιθώρια. Και τα πιλωτικά προγράμματα και αύξηση που ζητάμε κινδυνεύουν η κατάσταση είναι δραματική. Και επειδή το 2017, όπως θα πούμε και με τον συνάδελφο Σβέρπ ε, στην έκθεση εκτέλεσης του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, θα ε, ε, συζητηθεί το μέλλον των προγραμμάτων και η αναθεώρηση των προγραμμάτων, πρέπει να δώσουμε ένα στεναρό μήνυμα σε αυτό τον προπολογισμό, ο οποίος είναι και η διασταύρωση πολλών ευκαιριών. Για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο 2017 θα έχουμε τη νέα μεταρρύθμιση. Επομένως θα δούμε και τη διεύρυνση των συμμετοχόντων έχουμε τρει πόλει αντί για δύο ε, για πολιτιστικέ πρωτεύουσε. Επομένω, πρέπει κάπω να αντανακλώνται και όλα αυτά στον προπολογισμό. Θα ολοκληρώσω, μακρηγόρησα λίγο, αλλά να σα πω ότι αυτό το θέμα για μα είναι ζωτική σημασία σήμερα. Ευχαριστώ του ομιλητέ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σδρογεύσκη και του κοιόδη And <laughs> Και τώρα κάποιοι εξ ημών θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Όσοι δεν έχετε δουλειά, παρακαλώ να αποχωρήσετε.